Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο. Είμαι εντελώς κατά λάθο εδώ. Ε, είναι σαν να μπερδέψαμε τις καταχωρήσεις στο Μητρό. Λοιπόν, σε αυτό, αυτή την τεράστια αίθουσα θα ακούσουμε δύο εκθέσεις. Την πρώτη του κυρίου Κάρινς και α, ε, της κυρίας Κλέβα. Και οι δύο εισηγητές είναι εδώ και ξεκινώ με τον κύριο Κάρινς λόγω της ποιότητας του ακροατηρίου δεν είστε υποχρεωμένος να μιλάτε για πάνω από μισή ώρα βέβαια. Α, ο κύριος Κλούτ. Α, δεν υπάρχει διευμηνία στην γερμανική γλώσσα υποστηρίζει ο κύριος Σουκλούτε. Εντάξει. Λύθηκε το πρόβλημα, λέει στα γερμανικά ο κύριος ε, Πρόεδρος. Ο κύριος Κάριν, σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη. Εδώ και 7 λεπτά έπρεπε να είμαι στο κτίριο της Επιτροπής ε, γιατί ξέρετε ότι εμείς πήραμε την τελική επίσημη απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ για να συνδεθούμε με το ευρώ, για να ενταχθούμε συγγνώμη στο ευρώ και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα μείνω πάρα πολύ ώρα εδώ. Κύριε Γκοζές, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος και όχι μόνο για λίγο. Λοιπόν, τώρα θα κάνω όμως παρόλα αυτά την προβλεπόμενη σύντομη παρέμβασή μου. Να υπογραμμίσω ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όλοι μας, νομίζω, πάνω στο οποίο όλοι μας καλούμεθα να συμφωνήσουμε. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο χρειαζόμαστε στην Ευρώπη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις απασχόληση. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν σε αυτό. Εφόσον απαιτούνται λοιπόν οι επενδύσεις πρέπει να υπάρχει ένα ανεμπόδιστο τοπίο για να έρθουν οι επενδύσεις. Πολλές φορές δεν υπάρχει αυτή η ισονομία που απαιτείται και υπάρχουν ε, καταστάσεις οι οποίες από τους επενδυτές κρίνεται ότι παρεμποδίζουν ε, τις επενδύσεις. Και γι' αυτό ακριβώς λοιπόν και το θέμα της φοροδιαφυγής ε, είναι κάτι το οποίο παρεμποδίζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει μέσω της βελτίωσης των μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας. Το IMF, το ΔΝΤ, λέει ότι το 5% ε, του ΑΕΠ της Υπήρους μας είναι ε, παράνομο. Αν είναι αλήθεια αυτό, αν αληθεύει, είναι πραγματικά πολύ ψηλό το ποσοστό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα. Με την συγκεκριμένη οδηγία Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και οι τροπολογίες τις οποίες έχω εγώ καταθέσει θεωρώ ότι στην ουσία αποτελούν κάποια, κάποια σημεία επεξεργασίας, εκλέπτυνσης, αν θέλετε, κάποιων λεπτομεριών και όχι αμφισβήτησης της εκθέσεως. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Το πρώτο, αυτό το οποίο κατ' εμέ είναι και το πιο σημαντικό στα πλαίσια αυτής της, ε, της ε, οδηγίας είναι είναι το θέμα το ποιος θεωρείται σε κάθε περίπτωση αυτός ο οποίος ωφελείται και ποιος είναι ιδιοκτήτης ενός συγκεκριμένου σχήματος επενδυτικού είτε έχουμε να κάνουμε με το, με το φόρο τον οποίο κάποιος χρωστά, είτε ε, με την ε, μείωση των παρανόμως, ε, των παρανόμως διακινούμενων ποσών και ποιος ωφελείται από αυτά, το θέμα είναι ότι θα πρέπει οι ελεγκτικές αρχές να μπορούν να το ελέγξουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νομοθετικά χωρίς να έχουμε πάντα βέβαια το σύνολο ε, της εικόνας. Αλλά παρόλα αυτά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει ε, στα εταιρικά στοιχεία των επιχειρήσεων να καταγράφεται, να διευκρινίζεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Οι τράπεζες όταν ανοίγουν ένα λογαριασμό έχουν φυσικά τον κατάλογο των σημαντικών προσώπων της επιχείρησης, το ελέγχουν αυτό και θα βοηθούσε αν και τα μητρώα των επιχειρήσεων έπρεπε να έχουν αυτό το στοιχείο. Ε, θα πρέπει δηλαδή για να εγγραφεί μια επιχείρηση στα Μητρώα θα πρέπει να δώσει το κατάλογο των προσώπων που συμμετέχουν και ποιοι είναι τελικά οι πραγματικοί δικαιούχοι έτσι ώστε σε αυτά τα μητρώα να μπορούν να καταφνά προσφεύγουν οι αρχές όχι μόνο της συγκεκριμένης χώρας αλλά και άλλων χωρών. Οι ε, αρχές της Λετωνίας, σαν παράδειγμα, να μπορούν να δουν τι περιγράφει και τι περιέχει το πολωνικό μητρό εφόσον η εταιρεία αυτή ε, έχει την έδρα της εκεί, στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει λοιπόν α, α, αυτά να προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε μέσω της τροπολογίας 19. Νομίζω ότι έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και στην καταπολέμηση των παρανόμων εσόδων, από, των εσόδων μάλλον από παράνομες δραστηριότητες. Τώρα για την αξιολόγηση του κινδύνου και του επίπεδου κινδύνου. Έχει μεγάλη σημασία το ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να αξιολογεί τους κινδύνους για έκπληνση χρημάτων ή για ε, ε, φοροαποφυγή. Υπάρχει η τροπολογία 11 Υπάρχει η τροπολογία 11 που λέει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κίνδυνοι θα πρέπει να αξιολογούνται ανα επίπεδο σε επίπεδο χώρας σαν παράδειγμα ε, το κράτος μέλος ε, πρέπει να το ελέγχει αυτό και να έχει μία άποψη αλλά υπάρχει και η αντίστοιχη άποψη σε κοινοτικό επίπεδο. Και η ενημέρωση θα πρέπει να προέρχεται όχι μόνο από το εθνικό επίπεδο αλλά και από το κοινοτικό επίπεδο. Τώρα για την τροπολογία 24, νέες τεχνολογίες. Ε, την ε, επαφή κατά πρόσωπο ή όχι. Όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα όπως η ηλεκτρονική υπογραφή σαν παράδειγμα, ε, εδώ τίθεται, είναι το αντίστοιχο αν θέλετε με την φυσική παρουσία των μερών. Το θέμα δεν είναι να είναι κανείς υπέρ ή κατά της φυσικής παρουσίας, αλλά να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Τέλος, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με τις τροπολογίες αυτές και με την οδηγία αυτή, συναντήθηκα με αρκετούς εκπροσώπους της βιομηχανίας, με τα λεγόμενα λόμπις. Και είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκπρόσωπο, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Εταιριών που ασχολούνται με τα στοιχήματα υποδρόμου, τα υποδρομιακά στοιχήματα στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω ποια είναι η παράδοση στην Ιρλανδία, αλλά μου είπαν ότι στη χώρα αυτή μπορεί να κάνω λάθος. Υπάρχουν ε, τουλάχιστον 900 σημεία στα οποία μπορεί κανείς να πηγαίνει και να βάζει στοιχήματα, αλλά όλα αυτά γίνεται μόνο με ρευστό όλα πρέπει να γίνονται ε, πολύ γρήγορα με μηχανικό τρόπο και, και είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρει αυτούς που θέλουν να ξεπλύνουν έτσι και αλλιώς ε, χρήματα γιατί ε, τα έσοδα από, τις, από τα pounds τα οποία επενδύεις, από τις λίρες τις Ιρλανδικές που επενδύεις είναι πάρα πολύ περιορισμένα. και αυτό θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την ισχύ της συγκεκριμένης πρότασης. Αλλά μετά σκέφτηκα λίγο όπως σκέφτεται αυτός ο οποίος ξεπλένει χρήμα. 10% θα χρησιμοποιείται μόνο για να νομιμοποιήσει τα χρήματα του. Οπότε το 10% είναι πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι πληρώνουμε εμείς για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή. Ακόμα λοιπόν και για πάρα πολύ συγκεκριμένες ε, τέτοιες δραστηριότητες ε, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να ενσκύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαγράψει αυτή τη δραστηριότητα, αλλά να βρεθεί κάποιος τρόπος έτσι ο καταγραφής αυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία για να μπορεί κανείς να γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τα κέρδη τα οποία μπορεί να βγάλει από αυτό. Αυτά λοιπόν τώρα χοντρικά για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του ποσού μια συναλλαγή σε ρευστό που μπορεί να αμφισβητηθεί ή όχι, ιδιαίτερα στον τομέα των στοιχημάτων. Ίσως να μην ενδιαφέρονται άμεσα αυτοί που ξεπλένουν χρήμα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ίσως όμως και να ενδιαφέρονται, γιατί με ένα φόρο 10% ουσιαστικά αυτό ακούγεται ιδιαίτερα συμφέρον, δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ υψηλή η φορολογία. Ας μην λοιπόν καταστρέψουμε μια δραστηριότητα στην Ευρώπη λόγω της επιθυμίας μας να μειώσουμε το, το ξέπλυμα του χρήματος. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να διασφαλίσουμε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες έτσι ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους αλλά να μην διαγράψουμε την ίδια την ε, επιχειρηματική δραστηριότητα. Εγώ θα δω ε, τη συζήτηση αυτή που θα ακολουθήσει σε βίντεο, ένας από τους βοηθούς μου θα το φροντίσει και θα συνεργαστώ με τους κοιόδης συζητητές των υπολείπων ομάδων, αλλά όπως είπα πρέπει να αποχωρήσω. Ναι, ε, νομίζω ότι θα πάτε στους εορτασμούς για την είσοδο της Λετωνίας στην Ευρωζώνη. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εισηγητή του άλλου θέματος για τις διασταυρούμενες συνέπειες. Έχετε τον λόγο κυρία μου. Μετά την παρουσίαση της οδηγίας επιτρέψατε μου να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας παρουσιάσω το σχέδιο του τεχνικού μικρού αδελφού, το θέμα της μεταφοράς ε, κονδυλίων. Έχουμε τον ίδιο γενικό κανόνα. Ο κανονισμός προσπαθεί να δει την διαφάνεια ε, των εμβασμάτων, των μεταφορών χρημάτων διασενοριακά, ούτω ώστε οι διοκτικές αρχές να μπορούν να ανοιχνεύσουν, να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά τι γίνεται από εγκληματίες και από τρομοκράτες. Προσπαθούμε να έχουμε τις βασικές πληροφορίες των πληρωτών, των αποστολέων, ε, για να έχουν τις πληροφορίες αυτές οι διοκτικές αρχές ε, και να μπορούν να ανοιχνεύσουν εγκληματικές ενέργειες ε, και τα ίχνη τρομοκρατών. Ο στόχος είναι ο ίδιος, Έχουμε την, πρέπει να ε, συμμορφώνονται με τα διεθνή στάνταρτ, με τα διεθνή πρότυπα, ε, πρέπει να βρούμε την ανιχνεσιβότητα, την ιχνηλασιμότητα ε, των διαφόρων δράσεων και να συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα. Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν πέρσι τον Φεβρουάριο, η ΦΑΤΦΑ Νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να συνάδουν με τις αλλαγές των διεθνών προτύπων. Οι νέες απαιτήσει που έχουμε είναι ότι τόσο οι πληροφορίες ε, και όσο ε, οι πληροφορίες ε, για αυτόν που λαμβάνει την πληρωμή πρέπει να υπάρχουν και οι αρχές θα πρέπει να έχουν τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται. Επίσης ο άλλος συγητής ανέφερε αυτή την βάση κινδύνου, ε, πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να ενισχύσουμε μερικά από τα σημεία, τα υποκείμενα σημεία. Προτείνομαι να το κάνω αυτό συνδέοντας τη ρύθμιση με το παράρτημα της οδηγίας όπου προσδιορίζονται οι ε, παράγοντες υψηλού κινδύνου που θα αποτελέσουν δείκτες ή ενδείξεις για να μπορέσουμε ε, να οικοδομήσουμε αυτά τα μέτρα. Είναι σημαντικό να ε, έχουμε όχι μόνο ανεπαρκείς πληροφορίες, αλλά με την effective risk approach ε, να, έχουμε, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ε, μεταφορές αυτές ε, και να λάβουμε την, τα μέτρα που απαιτούνται. Αυτό ισχύει και για τις μεταφορές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε ήδη τέτοιες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές. Έχω εισαγάγει τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να περιλάβουμε. Ένα άλλο θέμα είναι ο διευκρινισμός ε, των ενδιαμέσων, ε, ε, των, αυτών, των παρόχων ενδιαμέσων υπηρεσιών, των ενδιαμέσων παρόχων υπηρεσιών. Είναι μια σύσταση της ΦΑΤΦ και νομίζω ότι η διαφορά υπάρχει και θα πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Οι δύο οντότητες δεν έχουν ίδια ε, ε, σχέση με τον πληρώνων και τον πληρωνόμενο, αυτόν που λαμβάνει την πληρωμή. Θα πρέπει να δούμε ε, ποιες πληροφορίες λείπουν και να υπάρχει στρατηγική παρακολούθηση που να εφαρμόζονται. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ρόλος και οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι οι ίδιες σχετικά με τους αρχικούς παρόχους υπηρεσιών Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει κάνει καλή εργασία ενισχύοντας το επίπεδο των κυρώσεων. Αυτό που με απασχολεί είναι η παρακολούθηση και η εκτέλεση, η πραγματοποίηση των κυρώσεων, κυρίως όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εναρμόνιση και θα ήθελα στα επόμενο έτος η Κομισιό να μας αναφέρει ξανά σχετικά με την εφαρμογή και την πραγματικότητα. Τι γίνεται στην πραγματικότητα Νομίζω ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των κρατών είναι κάτι το σημαντικό κυρίως όσον αφορά στις κυρώσεις. Επίσης νομίζω ότι έχουμε εδώ περιθώριο ελιγμού ε, για να μπορέσουμε να αρμονίσουμε τα δύο αυτά κείμενα ε, με την άλλα κείμενα, το CRD4 δηλαδή την ε, κεφαλαιακή επάρκεια 4 και θα πρέπει να στον τομέα της ε, καταπολέμησης του ξεκλίματος ε, χρήματος πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις κυρώσεις. Τελικά νομίζω ότι υπάρχει γενική κατανόηση. Με συγχωρείτε αλλά δεν έχω πλέον τη γαλλική μετάφραση. Α, έσβησε, έσβησε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει γενική κατανόηση ότι μπορεί να προκληθεί τεράστια ζημιά εάν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα δεν είναι παρκώς ε, προστατευμένα από καταχρήσεις εκ μέρους εγκληματικών ή τρομοκρατικών κύκλων. Θα πρέπει επίσης ε, να προσαρμόσουμε το ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο και οι εγκληματικές δραστηριότητες να μην αυξάνουν, να αυξήσουν τα προβλήματά μας και να μην είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές και θα απαντήσετε εναλλάξα. Ο κύριος Πέτερ Ζήμων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές ειλικρινά ε, για ε, την εισαγωγή τους με μεγάλη διαφάνεια και ειλικρίνεια. Να συμπληρώσω μερικά πράγματα. Ε, δεν χρειάζεται να συζητάμε εδώ επί της ουσίας για τη σημασία του νομοθετικού αυτού για ε, την αποτροπή χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος. Δύο δισεκατομμύρια δολάρια συμφώνησε να πληρώσει η HSBC στην Αμερική ε, για θέματα ξεπλήματος και τρομοκρατίας. Στην Ευρωπόλ επίσης βλέπουμε τέτοιους μηχανισμούς ξεπλήματος. Ε, ε, σφίγγουν οι έρευνες και στις επενδύσεις υποτιθέμενες για πράσινες επενδύσεις οικολογικές μέχρι και την Τράπεζα του Βατικανού. Έχει φτάσει αυτή η υπόθεση και χρειάζεται δράση. Συμφωνούμε ότι για να σταματήσει η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος, ποιο φυσικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται κανείς να μπορεί να κρύβεται πίσω από ε, και θολές κατασκευές. Ε, γι' αυτό ε, θα πρέπει να δούμε την έδρα διαφόρων ε, εταιριών, τα καταπιστεύματα να είναι όλοι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τους πραγματικούς δικαιούχου. Ε, προτείνει ο εισηγητή να προχωρούμε ακόμα περισσότερο στο εμπορικό μητρό, να συμπληρώνονται τα στοιχεία των δικαιούχων. Ε, αν θέλετε να προτείνω εγώ να κάνουμε ακόμα ένα βήμα. Για ποιο λόγο να μην μπορούμε να το ε, κάνουμε πανευρωπαϊκά ε, συντονισμένα, γιατί να το αφήσουμε στα χέρια των κρατών μελών. Ας πούμε το πεδίο εφαρμογής και την υποχρέωση αποκάλυψης ε, να ε, τα επεξεργαστούμε. Υπάρχουν ήδη οδηγίε για να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη ένα ελάχιστο ίση πληροφόρηση. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, τα τυχερά παιχνίδια που αναφέρθηκαν προηγουμένως και τον τζόγο και τα στοιχήματα. Η κυρία Κλέβα φώτισε τη μία πλευρά που χρειάζεται πιο σκληρή αντιμετώπιση να φωτίσω εγώ την άλλη. Ε, για να σκεφτούμε και άλλες εξαιρέσεις που ακόμα δεν έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως προς τον κίνδυνο, ας πούμε. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια της ε, ε, προσπάθειας αυτής να απλουστεύσουν τις υποχρεώσεις δήλωσης. θα πρέπει να το αξιολογεί ε, αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, και σε κάποιες περιπτώσεις να εξαιρούνται εντελώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα κρατικά λαχεία, το λότο στη Γερμανία. Δεν υπάρχει ούτε ο παραμικρός κίνδυνος επίθεσης ε, πάνω από 1000 ευρώ κέρδη ποτέ δεν καταβάλλονται σε μετρητά. Τα πρακτορία γνωρίζουν ότι όταν κερδίσεις πάνω από 1000 ευρώ δεν ξέρουν τα πρακτορία στοιχημάτων πόσο είναι το ποσό. Αυτό το ξέρει μόνο η εταιρεία στοιχημάτων και εμβάζει το ποσό στο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Μέχρι 999 καταβάλλονται σε μετρητά. Αφήστε δε που πάντα τίθεται το ερώτημα. Αναφέρθηκε επανειλημμένα. Ε, αν υπάρχει δυνατότητα ξεπλήματος χρήματος αγοράζοντας κάποιος ε, ένα ε, δελτίο που έχει κερδίσει παράνομα. Και ποιος παρακαλώ πολύ πουλάει ένα λότο που έχει κερδίσει νόμιμα ένα εκατομμύριο και μπορεί να πάει σε κάθε τράπεζα για να το πληρώσει για κάτι παραπάνω που τελικά και δεν θα μπορέσει ο ίδιος να δικαιολογήσει που τα βρήκε. Διότι έχει ξεφύγει από τον ε, νόμιμο διάβλο των κερδών και της διανομής. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος εκτίθεται σε ένα τέτοιο κίνδυνο και για ποιο λόγο. Για την εφαρμογή. Ορισμένοι συναδελφοί είπαν ότι η επιτυχία της εφαρμογής της οδηγίας ε, θα κριθεί από την ε, υλοποίηση, τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής ε, θα αναθεωρεί και θα εξετάζει την υλοποίηση στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι από τώρα μπορούμε να ελέγχουμε και να βοηθήσουμε για την επόμενη τετραετία. Μετά από τέσσερα χρόνια θα κάνει έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση. Θα μπορούσαμε ήδη από τώρα να προβληματιστούμε για το τι θα περιέχει αυτή, ε, τι θέλουμε να περιλαμβάνει μια τέτοια έκθεση, να υπάρχουν παράμετροι για τα κράτη-μέλη και να ξέρουν πού θα κριθούν, ποια είναι τα κριτήρια στα οποία θα μετρηθούν. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ. 15 μιλητές έχω προς το παρόν. Θα βάλω χρονόμετρο, δύο λεπτά έκαστος. Διότι στις 4 έρθει ο Υπουργός ε, Οικονομικών της Σλοβενίας. Κύριε Νίτρας, έχετε το λόγο. Βεβαίως θα περιοριστώ στο χρόνο, θα πω πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία είχα προβλέψει. Αλλά στον κύριο Σίμων μια παρατήρηση. Οι ρυθμίσεις που αφορούν το λότο ε, είναι ένα σύστημα, υπάρχουν σε πολλές χώρες, ένα σύστημα που δεν είναι και τόσο καθαρό, γιατί βλέπουμε εκεί τι κερδίθηκε, αλλά επειδή τα, τα άτομα δεν αναφέρονται προσωπικά, δεν βλέπουμε ποιοι έχασαν, βλέπουμε ποιοι κέρδισαν, ποιοι είναι οι κερδισμένοι, αλλά όχι ποιοι είναι οι χαμένοι. Όταν λοιπόν φτάνουμε ε, στα καζίνα, σε αριθμούς σημαντικούς, μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για το ξέπλυμα ε, χρήματος. Συμφωνώ γενικά με τα όσα είπαν οι συγητές, αλλά θα ήθελα να πω προς ποια κατεύθυνση θα ήθελα ε, να προσανατολίζεται η πρόταση, η ορισμός στο 217, τι Ποια είναι, ποιος είναι ο ορισμός εδώ, δεν είναι σαφής. Ποια είναι η συναλλαγή, εάν η συναλλαγή η οποία ήδη έχει αρχίσει από αυτόν που θα ωφεληθεί, μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ή όλοι ή όχι. Ε, καταλαβαίνω ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει να προσδιοριστεί καλύτερα η συναλλαγή μέσα στην Ένωση, αλλά θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια απλουστευμένη πληροφόρηση. Άρθρο 5, παράγραφος 1, θα ήθελα να την αναλύσω υπό το φως του άρθρου 4 μιλώντας για τους ε, προμηθευτές. Οι προμηθευτές δίνουν τον αριθμό του τιμολογίου ή έναν άλλο κωδικό αριθμό, αλλά δεν δίνουν τον τόπο κατοικίας. Εδώ μπορούμε, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μερικές δυσκολίες η τράπεζα δεν θα μπορεί πλέον να εξασφαλίσει την παρακολούθηση αυτών ε, των συναλλαγών, όπως θα είναι ε, δύσκολο να δούμε τις πηγές χρηματοδότησης ε, της τρομοκρατίας. Επίσης το κατόφλι των χιλίων ευρώ, δεν ξέρω, θα πρέπει οι τράπεζες πιστεύουν να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες για όλες τις συναλλαγές, όχι μόνο για τις συναλλαγές που ξεπερνούν ε, τα χίλια ευρώ. Το ίδιο πράγμα για τους ενδιάμεσους. Ακόμη και ε, κάτι άλλο. Ε, ως θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα των whistleblower που και να έχουμε μηχανισμούς που να επιτρέπουν την παρακολούθηση των συναλλαγών διότι υπάρχουν καταστάσεις όπου οι τράπεζες όχι μόνο δεν αποκαλύπτουν ε, τα δικήματα αλλά κατά κάποιο τρόπο συμμετέχουν σε αυτά τα δικήματα. Με συγχωρείτε που θα σας περιορίσω για την Άλντε η κυρία Ιντβελτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη διότι νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο των τροπολογιών δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα κάνω απλώς μια γενική παρατήρηση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε όλη την αιτιολόγηση πίσω από όλα αυτά. Έχουμε τους νέους ε, κανόνες FAGF αλλά θα πρέπει να δούμε ε, τι έχουν επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Αυτά οδηγούν οδηγούν σε περισσότερη ασφάλεια και ίσως ναι, αλλά θα ήθελα να έχω περισσότερες αποδείξεις Μερικοί είπαν ότι ε, έχουν κάποιο σκεπτικισμό για όλα αυτά. Νομίζω ότι μετά τα όσα μάθαμε τις πρόσφατες εβδομάδες για το βαθμό μέχρι του οποίου παρακολουθούνται οι πολίτες, νομίζω ότι θα έπρεπε να, είμαστε περισσότερο επικριτές, ε, περισσότερο σκεπτικιστές. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα απορρίψουμε εξ αρχής κάθε πρόταση. Θα ήθελα ε, να Έχω περισσότερες ε, αιτιολογήσεις. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν ένα βγνέο φόρτο γραφειοκρατικό ε, και επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών είναι σημαντικά. Πρέπει τα μέτρα αυτά να είναι απαραίτητα και να είναι αναλογικά. Αυτό απαιτεί ο νόμος. Εγώ φοβάμαι, παραδείγματος χάρη, ότι αν υποχρεώσουμε τις ε, εμπορικές επιχειρήσεις να συλλέγουν πληροφορίες για την αστυνομία, βρισκόμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Ε, είναι σαν να αναθέτουμε σε τρίτους ε, το έργο της αστυνομίας. Θα πρέπει να συλλέγουν οι επιχειρήσεις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για αυτές μόνο. Όταν ερχόμαστε στις λεπτομέρειες υπάρχουν μερικά ε, στοιχεία τα οποία δεν έχουν τη θέση τους σε μια νομική έκθεση ε, για την ε, κράτηση, διακράτηση των προσωπικών δεδομένων, η περίοδος, νομίζω ότι έχουμε τους νόμους, τους σχετικούς που ισχύουν. Δεν νομίζω ότι, ότι εμπίπτει στην εικόνα να προσδιορίσει τι είναι ύποπτο, τι είναι κίνδυνος. Νομίζω ότι αν ορισμένα στοιχεία δεν, έχουν, δεν είναι πλήρη, δεν θα πρέπει η ΕΚΟΝ να προσδιορίσει αν είναι ύποπτα τα στοιχεία αυτά ή επικίνδυνα. Θα ήθελα να τα εξετάσουμε όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να έχω περισσότερες βασικές αιτιολογίες γιατί θα πρέπει η ΦΑΤΦΑ να την, να την ακολουθούμε πιστά και τυφλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόρβαλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισήγητη για την γνωμοδότησή του. Αν και υπάρχουν σημεία όπου η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να βελτιωθεί η οδηγία αυτή όπως και άλλες καλύπτει έναν τομέα αφορούν δραστηριότητες όπως επίσης και τα υποδρομιακά στοιχήματα στην Ιρλανδία μέχρι και την ύπαρξη μηχανών για τυχερά παιχνίδια στη Φιλανδία. Πολλές φορές οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και περιπλέκει την κατάσταση. Από την άλλη πρέπει να εγγυηθούμε την ενότητα της ενιαίας αγοράς. Η πρόταση είναι να βελτιώσουμε ε, τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις εθνικές αρχές, χωρίς όμως αν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε επικαλύψεις και συγχύσεις αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε μαζί με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση ε, του εισηγητή για περιοδική αξιολόγηση θα δούμε αν θα πρέπει να γίνεται κάθε δύο ή τρία χρόνια. Πάντως νομίζω ότι η ανάλυση κινδύνων θα πρέπει να γίνεται στην αρχή της διαδικασίας για όλους και στο ίδιο επίπεδο. Ε, και μετά η αρμοδιότητα από το ευρωπαϊκό επίπεδο να πηγαίνει στο εθνικό επίπεδο ανάλογα με την περιοδικότητα που θα αποφασιστεί. έτσι ώστε και οι χώρες να μπορέσουν να ενισχύσουν τις δικές τους ελεγκτικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταβάρης από τους Πρασίνους δεν είναι εδώ, δεν ξέρω αν τον αντικαθιστά κάποιος. Κύριος Γκίγκολτ, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε την ώρα αυτή να δώσουμε το λόγο στη Γιούντι της Αρχεντίνη που είναι η συγγήτρια στην Επιτροπή Ελευθεριών και Συχνά το κάνουμε αυτό, δεν ξέρω πρόεδρε. Εντάξει, παίρνω εγώ το λόγο και αποφασίστε εσείς ποια είναι η σειρά. Εγώ που να ξέρω. Δική σας δουλειά είναι αυτή. Να μιλήσω εγώ τώρα ή όχι. Ναι, ναι, μιλήστε. Στο τέλος η εισηγήτρια της Επιτροπής Ελευθεριών γιατί θα μπορέσει να σχολιάσει όλες τις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Μιλήστε τώρα εσείς και με τα τελευταία κυρία Σαρχεντίνη. Μάλιστα. Εγώ προσέχω πάρα πολύ να μην μπαίνω ποτέ στα χωράφια της Λίμπε. Και ως ε, πράσινοι σεβόμαστε πολύ τις αρμοδιότητες των επιτροπών. Θα ήθελα λοιπόν να πω καταρχάς το εξής. Όλο αυτό το θέμα του ξεπλήματος ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι και οικονομικό ζήτημα και αυξανόμενο και ίσως δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητάμε έτσι γενικώ. Ε, υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού. Διαστρεβλώνονται πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα τμήμα της αγοράς που είναι νομοταγές και τηρεί τους κανόνες και ένα άλλο τμήμα της οικονομίας δεν τηρεί τους κανόνες, αυτό δεν έχει να κάνει με θεμητό ανταγωνισμό. Δεν μπαίνω καθόλου στα ποινικά ζητήματα. Αυτό είναι ίσως περισσότερο θέμα της Επιτροπής Ελευθεριών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα ε, ε, ε, οικονομικού εγκλήματος και μας αφορά αυτό, και φορολογικού δηλαδή, φοροαποφυγή ή αποφυγή διαφόρων κανόνων που διέπουν τις χρηματαγορές. Έχουμε λοιπόν σημαντικά ζητήματα και εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών. Αν δείτε και τους υπολογισμούς του μεγέθους, ο καθηγητής Σνάιντερ στο Λίντς έχει καταλήξει σε απίστευτα ε, νούμερα και στοιχεία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την παραοικονομία και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και από τη δική μας σκοπιά την οικονομική. Για την έκθεση αυτή καθ' αυτή να πω μερικά βασικά. Το ουσιαστικότερο για μένα, και εδώ ίσως συμφωνώ με τη Σοφία Νετβέλτ, είναι όχι να προσθέσουμε νέους κανόνες, αλλά να φροντίσουμε να εφαρμόζονται οι ισχύοντες και εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το ξεκαθαρίσει. Ότι δεν αρκεί να γράφουμε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να την ψηφίζουμε και μετά να διαφορούμε ε, για το εάν και κατά πόσο την εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις ε, που μπορεί κανείς να αμφισβητεί τη μεθοδολογία, αλλά είδαμε τι έγινε στην Κύπρο. Αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι λένε στα χαρτιά οι νόμοι. Όχι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία, οι τράπεζες, ε, αν είναι ε, νομοταγής και τηρεί τους κανόνες. Μπορούμε να ενισχύσουμε την έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή, ακριβώς χρησιμοποιώντας τις εποπτικές αρχές, για να βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε σκληρούς κανόνες και εφαρμόζονται κιόλας. Εγώ είμαι σκιώδης και μιλώ για δύο. Η πρόεδρος, α, θα μιλήσετε τέσσερα λεπτά, ωραία. Συνεχίστε, μιλώ για δύο. Εντάξει, δίκαιη ρύθμιση δεν είναι αυτή, ναι. Λοιπόν, τι έλεγα. Πέρα από αυτό, στην έκθεση δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο προτείνει ο εισηγητής να περιοριστεί ο υπολογισμός ε, των κυρώσεων ε, μόνο σε κάποιους στη θηγατρική. Δημιουργούν δηλαδή κάποιοι εικονικές εταιρείες θηγατρικές για να τους ρίχνουν τα πρόστιμα και να προστατεύονται οι ίδιοι από τις πιθανές κυρώσεις και πρόστιμα. Για μένα δεν έχει μεγάλο νόημα ε, αυτό. Επίσης, για ποιο λόγο η εφαρμογή που προτείνεται με ΑΙ πρέπει να είναι σε τέτοιο μακρύ χρονικό ορίζοντα. Και επίση θα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του τζόγου και το σωστό επίπεδο της διάκρισης. Το θέμα δεν είναι αν είναι ε, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου, αλλά αν υπάρχει κίνδυνος ξεπλήματος χρήματος. Αυτό θα πρέπει να είναι ο και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Ευχαριστώ. Τώρα θεωρητικά για άλλα τέσσερα λεπτά ο κύριος Τρέισεκ. <laughs> We will see. Thank you. Thank you, Madam uh, Ακούγοντας τη συζήτηση μέχρι τώρα, και γνωρίζοντας και τις θέσεις των σκιωδών εισηγητών, η θέση της ομάδας μου των συντηρητικών δεν διαφέρει και γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η κυρία Ιντβελτ είπε άλλωστε αυτά τα οποία θα ήθελα να πω κι εγώ, ιδιαίτερα την πρώτη μου παρουσίαση. Και επίσης κάτι από αυτά είπε και ο Γκίγκολντ. Να υπογραμμίσω όμως κάποια άλλα θέματα. Πρώτον, δεν θα πρέπει να εμείνουμε στο ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στις χρηματαγορές είναι ζαβολιάριδες, προσπαθούν να κάνουν απάτες και να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης οικονομικής κατάστασης, αυτό που θα μπορούσαμε να συστήσουμε είναι να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη κάτι που εγώ ε, θα ονόμαζα μέτρα διευκολυντικά της επιχειρηματικότητας και όχι βαρύτερες ρυθμίσεις γραφειοκρατικές οι οποίες μπορεί και να μην είναι απαραίτητες. Αντί να δημιουργήσουμε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ίσως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν οι ισχύουσες διατάξεις γίνονται αντικείμενο σεβασμού και αν εφαρμόζονται σωστά. Αυτά. Τώρα, δεύτερον, να πω και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κάριν στην εισαγωγική του παρατήρηση. Το 5% του συνολικού ΑΕΠ, του σφαιρικού ΑΕΠ που βασίζεται στους υπολογισμούς του ΝΙΤΑΦ είναι πραγματικά ένα τεράστιο ποσοστό. Αλλά είναι πραγματικά αληθινό εγώ νομίζω ότι είναι μια εκτίμηση, ένας υποτιθέμενος αριθμός. Θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Τώρα για τα εθνικά μητρώα. Η ενημέρωση στην καταπολέμηση του ξεπλήματος είναι κάτι το βασικό η θέση των εθνικών μητρώων, η δεκτικότητα των μητρώων, η προσβασιμότητά τους και το ποιος μπορεί να ενημερώνει και για τις διαμεθοριακές δραστηριότητες είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν περαιτέρω. Αλλά ακόμα και ο κύριος Κάριντς παραδέχτηκε ότι τα ενδιάμεσα μητρώα σε καμία περίπτωση δεν θα έλυναν το πρόβλημα. Οι νέες τεχνολογίες είναι το τελευταίο σημείο ζούμε στον 21ο αιώνα και δεν μπορούμε φυσικά να αποφύγουμε τις νέες τεχνολογίες και όσο περισσότερο εναρμονισμένη ε, είναι η διαδικασία τόσο περισσότερο οι νέες τεχνολογίες σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις ε, θα δημιουργήσουν νέες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις και ίσως εμπόδια. Ευχαριστώ. Θεωρητικά για άλλα τέσσερα λεπτά. Κλούτε. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να σύντομος υπόθηκαν ήδη πολλά και με κάλυψαν. Ε, θέλω να σας μιλήσω για μια άλλη πτυχή εγώ και να επικεντρωθώ εκεί. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε ότι το ξέπλυμα του χρήματος και η φορολογική απάτη όσο γίνεται θα πρέπει να αποφεύγονται. Πλην όμως θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Να μην το παρακάνουμε. Ναι, διατηρηθεί έτσι κάποια στοιχειώδης αναλογικότητα. Γιατί ακούμε συνέχεια καταγγελίες από πλευράς καταναλωτών και παράπονα ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτά τα θέματα ως πρόφαση για να αρνούνται στους πολίτες ε, να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό το λένε οι Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών επανειλημμένα ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην δώσουμε ένα επιχείρημα στα χέρια των τραπεζών και να ανοίγει μια πόρτα για να αυθαιρετούν. Δύο παραδείγματα έχω τα οποία αναφέρουν πάντα οι ενώσει καταναλωτών. Από τη Μεγάλη Βρετανία είναι το ένα πρόβλημα. Εκεί επιμένουν οι τράπεζες ότι κάποιος που θέλει να έχει ε, τραπεζικό λογαριασμό στη Βρετανία θα πρέπει να έχει και διεύθυνση κατοικία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι αυτό είναι προβληματικό, το γνωρίζει και θα πρέπει να κοιτάξει ε, ε, τι θα κάνει για πανευρωπαϊκούς κανόνες για το ξέπλυμα. Αλλιώ δεν λειτουργεί εσωτερική αγορά απλούστατα. Δηλαδή όταν έχεις μία εσωτερική αγορά δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις κάπως περίεργες και εμπόδια να δημιουργούνται ή να ορθώνονται. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να προσέξουμε, ε, μας το λένε επίσης οι καταναλωτές, ενώ του στη Γαλλία εν μέρη έχουν εμφανιστεί αυθαιρεσίες από τράπεζες και πάλι που λέγουν ότι είναι κατά του ξεπλήματος και συλλέγουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των πελατών και τα χρησιμοποιούν για σκοπούς διαφήμισης. Δεν το έχω δει προσωπικά, το έχω ακούσει από ενώσεις καταναλωτών. Ε, και αυτό είναι αυθαιρεσία. Τι δουλειά έχει εδώ το ξέπλυμα. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν σε αυτό το κανονισμό να μην υπάρχουν παραθυράκια για ε, καταχρήσεις και να διατηρηθεί μια στοιχειώδης αναλογικότητα, όπως είπα. Αυτά δεν θέλω να πω πολλά παραπάνω. Ένα τελευταίο σχόλιο, καταληκτικό. Συζητούμε πάντα με θέματα συμφωνιών, ελευθέρων συναλλαγών, ε, ε, ασχολούμαστε. Και ακριβώς, αν θέλουμε να αποτρέψουμε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, να έχουμε πιο σαφείς κανόνες σε αυτές τις συμφωνίες. Κολομβία, Περού, θυμίζω, δεν έχει μεγάλο νόημα μεταξύ μας να συνεννοούμαστε πώς θα αποφύγουμε το ξέπλυμα, ενώ σε συμφωνίες με τρίτες χώρες του κόσμου ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα ορθάνυχτα για το ελεύθερο ξέπλυμα. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Yes, I've had some interesting debate. Ναι, ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, έτσι μου λένε. Νομίζω θα πρέπει να δώσω τον λόγο στη Τζούζη της Αργεντίνη και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και ο υπουργό είναι εδώ ε, για την, ε, το επόμενο τμήμα της συνεδρίασης. Αλλά δεν θα υπάρχει χρόνο στο τέλος ε, για τον εισηγητή, η Τζούντιθ και μετά η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η δική σας παρατήρηση ότι έπρεπε ότι να, να δώσετε πάρα πολλά στοιχεία όταν χρειάστηκε να ανοίξετε ένα λογαριασμό είναι ένα στοιχείο κλειδί για αυτή τη συζήτηση πολλά έγγραφα. Νομίζω ότι η ΛΥΜΠΕ και η ΕΚΟΝ ε, θα έχουν αρμοδιότητα ε, για το άρθρο 51 και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί μετά το θέρος. Χαίρομαι που ε, θα είμαι μαζί σας για να συζητήσω αυτή την οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά θα αρχίσω με το βασικό θέμα για την Επιτροπή Οίκων που είναι η ε, το να περιλάβουμε ε, τα φορολογικά αδικήματα σε αυτό το κείμενα. Δεν υπάρχει ένας ορισμός των φορολογικών αδικημάτων. Αν αφήσουμε τον ορισμό στα, 8, ε, στα 28 μέλη, θα έχουμε ένα νομοθέτημα χρήσιμο που θα μπορεί να καταπολεμήσει τα φορολογικά αδικήματα, ο συνάδελφος Γκίγκλτ λέει, που θα μπορούμε να εφαρμόσουμε την, ε, την νομοθεσία που έχουμε εδώ επιτάπητος, αν δεν διευκρινίσουμε κάτι για το τι είναι ένα φορολογικό αδίκημα, είναι ένα αδίκημα, είναι ένα έγκλημα, ε, σε πολλές χώρες ε, η αποφυγή των φόρων δεν θεωρείται αδίκημα, αλλά σαν μέτρο διοικητικό τότε δεν θα έχουμε τίποτα. Θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την διαφορά ανάμεσα στην φορολογική απάτη και στο φορολογικό αδίκημα. Η φορολογική απάτη έχει ήδη προσδιοριστεί, το αδίκημα όχι. Το G8 ζήτησε δράση από τα κράτη-μέλη ε, για τα φορολογικά αδικήματα, αλλά ε, ζήτησε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ε, για την φοροδιαφυγή και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος, η καλύτερη διέξοδος αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο αυτό έχει ε, την ευθύνη να προσδιορίσει τι είναι το φορολογικό αδίκημα. Δεν είδα τον εισήγητη τη ΕΚΟΝ να το πράττει. Ε, θα ήθελα ε, και ζητώ από τους σκιώδεις να εξετάσουν το θέμα αυτό. Μετά όταν ε, προσπαθούμε να δούμε τι είναι οι κίνδυνοι και ποιος προσδιορίζει τους κινδύνους. Έχουμε την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Τραπεζών, έχουμε την Europol, έχουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλιών και Συντάξεων, έχουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. ποιος είναι αυτός που ελέγχει όλες αυτές τα όργανα, την Ευρωπαϊκή Αρχή των Τραπεζών και κυρίως την Ευρωπόλ εμείς βασίζουμε την καταπολέμηση σε πληροφορίες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Πώς εμείς ως ευρωβουλευτές, ως εκπρόσωποι ε, του λαού ξέρουμε ότι κάνουμε τα σωστά πράγματα. Η κυρία Ινφέλντ ε, και άλλος σκιώδης εδώ ανέφεραν το θέμα της προστασίας δεδομένων και του ξεπλήματος και είναι δικό μας καθήκον να έχουμε να το καταστήσουμε αυτό ένα εργαλείο ε, χρήσιμο κατά της, ε, του ξεπλήματος αλλά ε, και της φοροδιαφυγής και των φορολογικών αδικημάτων. Δεν ξέρω αν ε, δεν, ε, δεν ε, περιλαμβάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα που θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την νομοθεσία, με τι θα πρέπει να συμμορφώνεται, με το, ως προς το ξέπλυμα ή ως προς την προστασία δεδομένων. Νομίζω ότι οι πληροφορίες που έχει έκον δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούμε στα κράτη να έχουμε τις πληροφορίες που έχουν οι αστυνομίες. Ε, πολλοί σε μερικές χώρες ε, υπερέχει αστυνομία, σε άλλες όχι. Θα πρέπει να, ε, να αφήσουμε αυτό το θέμα της προστασίας δεδομένων, τελειώς θα έχουμε ένα σωρό και προσφυγές και δεν θα έχουμε καλή νομοθεσία κατά πολέμησης του ε, ξεπλήματος. Και το τελευταίο μου σημείο, κυρία Πρόεδρε και θα κλείσω, πώς θα το κάνουμε αυτό αποτελεσματικά όταν υπάρχουν 28 κράτη-μέλη με 28 συστήματα, καθεστώτα διαφορετικά, όπου κάθε τράπεζα, ε, κάθε οργάνωση παιχνιδιών ε, θα έχει ε, την δική του ιδέα του τι είναι ένας κίνδυνος και αν ο κίνδυνος είναι κίνδυνος σε μια χώρα και όχι σε μια άλλη χώρα, πώς θα βεβαιωθούμε ότι διασυνεργειακά αντιμετωπίζουμε το ξέπλυμα χρήματος και την φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε επιτάπητος δεν είναι αρκετό και θα πρέπει να εργαστούμε για να γίνει επαρκές. Τελευταία παρατήρηση, τελευταία, τελευταία, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι... Ε, ε, λυπούμε, λυπούμε. Δεν μ' αρέσουν αυτέ οι παρατηρήσει και είναι πάντα οι πράσινοι που μου κάνουν. είναι πάντα οι πράσινοι που μου κάνουν τέτοιε παρατηρήσει. Η προσέγγιση που βασίζεται στο κίνδυνο. Όλοι μου λένε ότι η προσέγγιση αυτή είναι καλύτερη. Είμαι έτοιμη να το πιστέψω, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιος ερευνά τους κινδύνους και θα ήθελα να ξέρω ότι αν ακόμα και η προσέγγιση αυτή η βάση κινδύνου βασίζεται σε κανόνες. Δεν μπορεί κανείς να εργαστεί χωρίς να ξέρει τον κανόνα, το κατόφλι, το κατώτατο όριο, το ποσό ε, των, ε, των λογαριασμών που ανοίγουν ή που κλείνουν. Νομίζω ότι είναι profiling αυτή η προσέγγιση και το profiling, τα προφίλ, είναι κάτι για τα οποία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, Τώρα δεν έχουμε ούτε χρόνο για την Επιτροπή, διότι έχω εδώ τον Υπουργό. Έχω δύο λεπτά για την Κομισιό. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, αλλά συγητής της ΛΥΜΠΕ πήρε το χρόνο σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και ευθύ στο πρώτο σημείο σχετικά με την σημασία του ξεπλήματος χρήματος και ξέρω ότι υπάρχουν ερωτήματα ε, για τις αποδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία, η προσέγγιση της ΦΑΤΦΑ ε, με τα διεθνή πρότυπα. Νομίζω ότι πρόκειται για έναν δύσκολο τομέα για να μπορούμε να αξιολογήσουμε όλο τον αντίκτυπο και όλο το σύστημα. Όλο ο τρόπος να εξετάσουμε όλο αυτό το θέμα είναι να διερωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα ισχύων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε εδώ κανόνες, κανόνες με αναλογικότητα για να βεβαιωθούμε ότι δεν πρέπει να επηρεάζουμε όλες οι επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο, διότι λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές και ορισμένες επιχειρήσεις ε, ε, τοποθετούνται διαφορετικά σε σχέση με τους κανόνες. Ε, σχετικά με τα φορολογικά δεν είμαστε αντίθετοι ε, με τα μητρώα επιχειρήσεων αλλά υιοθετήσαμε εδώ την προσέγγιση να συγκεντρωθούμε στην πηγή των πληροφοριών ε, και να θεωρούμε και να έχουμε τις πληροφορίες ως τον ετών πιο εγκαίρος. Οι επιχειρήσεις νομίζω πρέπει να έχουν τις πληροφορίες. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση ως προς τα τυχερά παιχνίδια. Έχουμε εδώ μια προσέγγιση βασική κινδύνου σε σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους και τον τομέα των παιχνιδιών. Έχουμε μια προσέγγιση με ευρύ ορισμό, αλλά επιτρέπει κάποια δυνατότητα ευελιξίας, ούτως ώστε να αξιολογούνται οι κίνδυνοι διαφορετικά στους διάφορους τομείς των παιχνιδιών ως προς την αποτελεσματικότητα των κανόνων θα πρέπει να επισύρουμε την προσοχή πάνω στην στο ευρύ διαδικασία που υπάρχει για την έλεγχο της αποτελεσματικότητας με την Task Force, η νέα προσέγγιση της ΦΑΤ θα βασίζεται περισσότερο στην αποτελεσματικότητα. Σε σχέση με την προστασία δεδομένων, έχουμε συνειδητά κάνει μια επιλογή να περιορίσουμε τον αριθμό ε, των κανόνων για την προστασία δεδομένων στην οδηγία. Η οδηγία κατά πολέμηση του ξεπλήματος είναι μέσα στο πλαίσιο το γενικότερο της προστασίας των δεδομένων. Είναι μια προσέγγιση που αναπτύξαμε κατόπιν διαβουλεύσεως με συναδέλφους ε, της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και του ε, επόπτη των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την ευχή του εισηγητή να υπάρχει προσέγγιση βάση κινδύνων ε, με ορισμό σε αυτήν, αυτήν την οδηγία κατανοούμε ότι υπάρχει κάποια ασάφεια. Θα επισύρουμε την προσοχή πάνω στο γεγονός όμως ότι έχει γίνει σημαντική εργασία όταν ο πρώτος κανονισμός εκπονήθηκε από τις εθνικές τραπεζικές αρχές, από τον Ευρωπαίο Επόπτη, που έχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ρόλο των ενδιαμέσων. Υπάρχει, είναι διαφορετικός ο ρόλος για αυτόν που πληρώνει, αυτόν που λαμβάνει την πληρωμή. Θα εξετάσουμε τις προτάσεις και τελικά το θέμα του ε, ναι ή όχι, το ευρωπαϊκό σύστημα, το ενδοευρωπαϊκό είναι ένα το οποίο θα είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθεί. Δεν το πιστεύουμε. Μπορεί να εποπτευθεί με την ε, ε, μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλές λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζουμε ότι τα κράτη-μέλη και ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση που έχει επίσης υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τέσσερα λεπτά και 35, εν πάση περιπτώσει θα καταφέραμε. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα ποια θα είναι η διαδικασία, δεν δίναμε. Κάποια στιγμή θα υπάρξει προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ή μπορεί να ξανανοίξει η προθεσμία για μια νέα έκθεση. Προς το παρόν έχουμε 18 τίνος 18 Ιουλίου Ενδιαφέρουσα ημερομηνία είναι αυτή. Μέχρι τι 18 Εβδόμου έχετε να κάνετε τροπολογίες. Εκτός αν υπάρξει διαφορετική ενδολή. Σας ευχαριστώ πολύ και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα τη ημέρης τη διάταξη, που είναι οικονομικός διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Οικονομικών της Σλοβενίας. Uh, λοιπόν, δύο σελίδες σημειώσεις έχω, δεν πρόκειται να τις διαβάσω, μην ανησυχείτε. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον Υπουργό Οικονομικών της Σλοβενίας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και τον οικονομικό διάλογο. Πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση. Θέλω να σας ενημερώσω ότι εκτός από τον παρόντα οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τη Σλοβενία σήμερα, έχουμε Είχα πριν από λίγες εβδομάδες αποστείλει επιστολή και προσκλήσει και σε άλλα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στο διάλογο. Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και Λουξεμβούργο είναι οι χώρε αυτές και περιμένω ακόμα επιβεβαίωση. Και θα σας ε, τηρώ ενήμερους βεβαίως ε, εν ευθέτω χρόνο. Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα και Λουξεμβούργο. Έχουν γίνει επαφές αλλά δεν έχουμε λάβει επιβεβαίωση. Από την Πορτογαλία καμία απάντηση. Και στο μεταξύ έχει αλλάξει και ο Υπουργό Οικονομικών. Μάλλον θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Και νέα πρόσκληση πρέπει να στείλω. Παρακαλώ όλα τα κράτη-μέλη να καταβάλουν ε, προσπάθεια να έρχονται στον οικονομικό διάλογο για να γίνεται μια γνήσια ουσιαστική ευρωπαϊκή συζήτηση για την πολιτική. Θα δώσω όσοι ήθιστε το λόγο στον Υπουργό Uh, το πολύ 10 λεπτά μπορείτε κύριε Υπουργέ να τα ε, καταφέρετε. Και μετά η ε, έρωτα ερωταποκρίσεις σε χρονοθυρίδες 5 λεπτών. Και ελπίζω να το τηρείτε. Και να μην τρώει το πεντάλεπτο ο εκάστοτε βουλευτής με την ερώτησή του και δεν έχετε χρόνο να απαντάτε. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ με μεγάλη μου χαρά αποδέχομαι την πρόσκληση και έρχομαι να σας μιλήσω για τον οικονομικό διάλογο και την οικονομική μας πολιτική. Είχα στην αρχή σκεφτεί να κάνω την εισαγωγή αυτή για την οικονομική πολιτική βασιζόμενο σε τρία σημεία. Να σας παρουσιάσω κάπως την οικονομική κατάσταση σήμερα στη Σλοβενία. Επίσης, ε, τις δραστηριότητες ε, στο οικονομικό πεδίο και μετά το δεύτερο πυλώνα κάποια σημεία που σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν και σας στη δουλειά σας. Πώς πάει η οικονομική κατάσταση στη Σλοβενία. Μετά από πέντε χρόνια αργής ανάπτυξης, που καμιά φορά δεν ήταν καν ανάπτυξη, αλλά ήταν στασιμότητα, μέχρι και ύφεση, Τώρα θα πρέπει να δράσουμε ε, ταχαίως και το γνωρίζουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε χαμηλό χρέος, 55% του ΟΕΠ, αλλά αυξήθηκε σημαντικά και γρήγορα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία έτη. Και το μοναδιαίο κόστος εργασίας δεν έχει αυξηθεί, ε, είναι στάσιμο και έχει αρχίσει να αυξάνεται στην αρχή της περίοδου. Δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα διαρθωτική προσαρμογή στην κρίση. Παρ' όλα αυτά, ε, είναι υγιή τα μακροοικονομικά μας ε, βασικά. Στα νοικοκυριά, ας πούμε, έχουμε τη χαμηλότερη ιδιωτική χρέωση στην Ευρώπη σχεδόν και το δημόσιο χρέος είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρώπης. Από την άλλη φορά, ε, από την άλλη πλευρά, συγγνώμη, έχουμε στις επιχειρήσεις ανισορροπίες. Είναι πολύ ψηλή η χρέωση των εταιριών και αυτό φαίνεται και στους ισολογισμούς των ιδίων των εταιριών αλλά και των τραπεζών. Και αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και ε, κάθε φορά που χαράσουμε οικονομική πολιτική. Ένα δεύτερο στοιχείο. Αν δείτε την τελευταία πενταετία, δεν ελήφθη αποτελεσματική πολιτική. Ε, έχουμε κάποιες ελλείψεις θεσμικές και καθυστερήσεις που πρέπει να καλύψουμε. Οπότε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ταχαίως και να προσαρμοστούμε ε, ορθώς στην οικονομική κρίση. Κάνοντας μια ανασκόπηση όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει κάποιες δράσεις στο παρελθόν, μεταρρύθμιση των συντάξεων, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και η εξυγίαση ε, του προϋπολογισμού άρχισε να εφαρμόζεται. Αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί. Έχουμε λοιπόν ε, ε, μια οικονομική πολιτική που βασίζεται σε τρεις πυλώνες πρώτος πυλώνας, πώς θα αλλάξει η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Καλωσορίζουμε την ε, νομοθεσία ε, για τα δημοψηφίσματα. Στο παρελθόν πολλές αποφάσεις ε, εμποδίστηκαν από δημοψηφίσματα, οπότε θα αλλάξουμε. Αλλάξαμε το Μάιο το Σύνταγμα και αυξήσαμε το κατόφλι που χρειάζεται για να διεξαχθεί δημοψήφισμα, οπότε είναι πιο ομαλή η νομοθεσία ε, των ε, μεταρρυθμίσεων. Κάτι που θα ήθελα να σας αναφέρω για το σύστημα ψηφοφοριών στη Σλοβενία. Έχουμε πολλά κοινοβουλευτικά κόμματα με μεγάλο συνασπισμό στην κυβέρνηση και είναι ασταθής. Το έχουμε δει στο παρελθόν η πολιτική σκηνή. Και αν θέλουμε να έχουμε λίγο πιο γερή οικονομική πολιτική και διαρκή, χρειάζεται πιο σταθερή κυβέρνηση κάθε φορά. Ένα επόμενο στοιχείο ε, των αποφάσεων είναι η οικονομική διακυβέρνηση. Στη Σλοβενία δεν είναι εξαιρετική, μάλλον το αντίθετο. Ε, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, δικούμε τις επιχειρήσεις μας. Όλα αυτά ε, ως οικονομικές αποφάσεις και διαδικασίες ε, είναι αλληλένδετα. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα της οικονομικής πολιτικής είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας. Μετά από μία πενταετία ύφεση θα πρέπει να εστιάσουμε πλέον στην ε, τόνωση της ανάπτυξης από τη μια και την εξηγήση του προπολογισμού από την άλλη. Θα σας μιλήσω περισσότερο στη συνέχεια γι' αυτά. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας είναι ουσιαστικά ο πυλώνας στον οποίο ε, εστιάζουμε πραγματικά πολύ βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να δράσουμε ταχαίως και αποτελεσματικώς έτσι ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε από εκεί και πέρα τα μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει ένα προγραμματισμό μακροπρόθεσμο για μεταρρυθμίσεις εάν παλεύει και αγωνίζεται να κανονίσει την καθημερινότητα και τα βραχυπρόθεσμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη στο Δυναικές, με μια οικονομία ε, ανταγωνιστική και με όρους που να ε, ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, να έχουμε ένα σύστημα θεσμικό που να λειτουργεί, να είναι ο δημόσιος τομέας ε, πιο περιορισμένος και πιο αποτελεσματικός και να βελτιωθεί και ε, το περιβάλλον αλλά και ο τομέας της υγείας και της περίθαλψης. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το δεύτερο πυλώνα. Έχουμε οικονομικές προτεραιότητες της εξής. Πρώτον, η ε, τόνωση της ανάπτυξης και πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό. το ισοζύγιο πληρωμών Και οι ισολογισμοί των τραπεζών ε, είναι προβληματικοί και δεν τους ε, επιτρέπουν ούτε να δανείζονται από τις αγορές, ούτε να δανείζουν ε, στις επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια μόχλευση λοιπόν να αρχίσουμε από τις αποκρατικοποιήσεις τραπεζών και μεγάλων κρατικών εταιριών ιδιωτικοποίηση και επίσης και ευραχυπρόθεσμα χρειάζεται κάποια βελτίωση στη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Ως προς το χρέος, Μάλλον ε, ε, έχουμε δημιουργήσει μια bad bank που θα αναλάβει το κακό χρέος που ήδη λειτουργεί. Η σχετική νόμη είναι στο νόμο παρασκευαστικό σχέδιο. Έχουμε συνεργαστεί με διεθνή ιδρύματα, η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης και Έχουμε εκλέξει και τους διευθυντές, εκτελεστικό και μη διευθυντή, με διεθνή εμπειρία. Και με εμπειρογνώμονες γενικότερα και τώρα είμαστε έτοιμοι για να ε, μεταφέρουμε κάποια στοιχεία του ενεργητικού στην Bad Bank αυτή. Ε, τις ε, ε, δοκιμασίες αντοχής, τα stress test επίσης θα πρέπει να κάνουμε και να μας δοθεί ε, η πλήρης άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Ε, ως προς τις ιδιωτικοποίησεις, αυτές βαίνουν παράλληλα. Έχουμε καταρτήσει ένα πρώτο κατάλογο εταιριών, 15 τον αριθμό, που επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθούν. Ε, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του Κοινοβουλίου βέβαια ως προς αυτό να εγκριθεί ο κατάλογος των 15 εταιριών που προορίζονται για ιδιωτικοποίηση. Έχουμε και ένα κατάλογο υποψηφίων πριν από ένα μήνα περίπου. Εγκρίθηκε ε, πριν από δύο εβδομάδες από το Κοινοβούλιο και τώρα θα αρχίσουμε να περνούμε στην υλοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουμε και το καθεστώς ε, της εταιρείας ε, που ασχολείται με τις ιδιωτικοποιήσεις. Ε, το φθινόπωρο, περί τα μέσα, θα έχουμε την πλήρη στρατηγική για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και ποιες εταιρείε κρατικές θα πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν οριστικά ή ποιες δεν πρόκειται. Η δεύτερη οικονομική προτεραιότητα είναι η εξυγίανση ε, του προϋπολογισμού των δημοσίων οικονομικών μας. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε ε, στην προσπάθεια της μείωσης του ελλείμματος. Ξέρετε ότι η Σλοβενία είναι μικρή και ανοιχτή οικονομία ε, είναι πολύ σημαντική να είναι ανταγωνιστική για να είναι και βιώσιμη ε, στο Δίνεκες, ε, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις δαπάνες και λιγότερο στα έσοδα. Σε γενικές γραμμές έχουμε μέτρα της τάξης του 1 δις, που είναι το 3% περίπου του ΑΕΠ μας. Αυτά τα μέτρα ε, ε, είναι στα δύο τρίτα από την πλευρά των δαπανών και στο 1 τρίτο από την πλευρά των εσόδων. Και θα πρέπει να εφαρμοστούν φέτος και αρχές του επομένου έτους. Η δική μας φιλοδοξία ουσιαστικά ήταν να τα εγκρίνουμε φέτος, ανεξαρτήτως ε, αποτελέσματος, αν θα απέδιδαν ήδη από το 2013 το 2014, για να προχωρήσουμε πλήρως αυτό το δρόμο της εξυγίασης των δημοσίων οικονομικών. Ένας ακόμα στόχος που έχουμε ε, είναι το χρέος. Είμαστε χώρα με χαμηλό χρέος, 55% του ΑΕΠ. Και ξέρουμε ότι για να έρθει η ανάπτυξη, να ε, υπάρξει αναδιάρθρωση και μεταρρυθμίσεις, για να γίνουν όλα αυτά θα αυξηθεί το χρέος μας, αλλά θέλουμε, ε, αφού ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, να το μειώσουμε ξανά και γι' αυτό ποντάρουμε και στην ιδιωτικοποίηση. Αυτά εισαγωγικά για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες και στη συνέχεια μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις αν χρειάζεται και εξηγήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Γκοζές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στη συνάντησή μας. Παρότι είναι μεγάλη αίθουσα, νομίζω ότι έχουμε μια καλή αίσθηση επικοινωνίας. Ε, εσείς είπατε, δώσατε κάποια στοιχεία, αλλά είπατε ότι περιμένετε και τις ερωτήσει, γιατί αυτά τα οποία μας είπατε μέχρι τώρα, ιδιαίτερα για την κατάσταση των πιστοτικών ιδρυμάτων και την δυνατότητα βοήθειας ε, ανάκαμψης των τραπεζών και το θέμα της υπερχρέωσης, ε, δεν μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία. Μπορείτε με λίγο πιο πιστικό τρόπο να μας πείτε ε, με ποιους τρόπους θα αντιμετωπίσετε θέματα των τραπεζών και κατά συνέπεια και το θέμα του χρέους. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Σχετικά με τις τράπεζες και το θέμα της ανάκαμψης των τραπεζών είναι το κέντρο θα έλεγα της οικονομικής μας πολιτικής. Εμείς θελήσαμε να το αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν και γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια bad bank. Ασχολούμεθα με το θέμα αυτό από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, Αύγουστο, με την προηγούμενη κυβέρνηση και η βασική ιδέα είναι από τη μία να δημιουργήσουμε αυτήν την τράπεζα η οποία θα κατέχεται 100% από το κράτος. Μια τράπεζα χρεών η οποία θα έχει σαν στόχο να επιτρέψει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να αγοράσει στοιχεία από τις τράπεζες αυτές και ομόλογα τα οποία θα εκδίδουν οι τράπεζες αυτές και για τα οποία θα δίδει εγγύηση το κράτος ή να δίδει εγγυήσεις επίσης για κάποιο είδους εκδόσεις από πλευράς άλλων τραπεζών. Δημιουργούμε το νομικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για να γίνει κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να περάσουμε την νομοθετική ρύθμιση μέσα από το Κοινοβούλιο. Δημιουργήθηκε, δημιουργήσαμε και ένα δημοψήφισμα. Τώρα τα πράγματα υπάρχουν, έχουν αλλάξει, υπάρχουν κάποιες μικρές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν Τρία πράγματα πρέπει να διευκρινίσω εδώ. Πρώτον, αυτή η εταιρεία bad bank, η κακή τράπεζα σε εισαγωγικά, θα πρέπει να ανήκει απολύτως στο κράτος. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και από τον ιδιωτικό τομέα, όχι ίσως για το πρώτο κομμάτι, για την πρώτη φάση, αλλά όταν διευκρινιστούν οι κίνδυνοι θα υπάρξει κάποια όρεξη θα έλεγα από τον ιδιωτικό τομέα για την ιδιοκτησία της συγκεκριμένης αυτής τράπεζας. Έχει σημασία να μειώσουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση το ποσοστό του κράτους. Είδαμε τι έγινε στην Ιρλανδία και την Ισπανία, 49% το ποσοστό του κράτους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορείς να αφαιρέσεις τα ποσά αυτά από το δημόσιο χρέος και να παρουσιάσεις τα, τα θέματα που αφορούν την κατάσταση των δημοσιονομικών με διαφορετικό τρόπο, με καλύτερο τρόπο. Ε, θα πρέπει να αλλάξει επίσης και ο νόμος ε, για τη διάρκεια αυτής της τράπεζας. Ε, πέντε χρόνια είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα όταν θέλει κανείς να αποεπενδύσει κάποια αγαθά, κάποια είδη ή κάποια προϊόντα, πέντε χρόνια είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει με νομική ρύθμιση να παραταθεί. Και τέλος, υπάρχει... Ε, of, ε, of 10%. Κάτι το οποίο θα κάνει ελκυστική νομίζω την προσπάθεια αυτή σε έφθετο χρόνο. Λοιπόν, έχουμε τον νόμο, έχουμε το πλαίσιο, υπάρχει διαχειριστική ομάδα. Θα υπάρξει και δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει και το πόσο υπόλογη θα είναι η διοίκηση της τράπεζας αυτής και μόλις πάρουμε το πράσινο φως και από τη Γενική Διεύθυνση την αρμόδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προχωρήσουμε. Θα πρέπει να μας δώσει την αδειά η αρμόδια Γενική Διεύθυνση γιατί υπάρχουν θέματα που άπτονται των κρατικών βοηθειών. Και αυτό θα μας βοηθήσει ε, για την ανακεφαλαίωση των υπολείπων τραπεζών και σε αυτή τη φάση αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του κράτους λόγω ακριβώς των συνθήκων που επικρατούν στις αγορές μου. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε το πράσινο φως, εν πάση Αυτά. Το αρχικό μας πρόγραμμα ήταν να υπάρξει μεταφορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να ξεκινήσουμε με το πρώτο πακέτο πριν το τέλος του Ιουνίου, να γίνει αξιολόγηση τον Ιούλιο, για να περάσουμε στο επόμενο, ε, θα έλεγα, στο επόμενο σχολικό έτος, ξεκαθαρίζοντας τις σλοβενικές τράπεζες. Ελπίζω να ήμουν ε, επαρκή στην απάντησή μου. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση από την κυρία Κλάβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό λοιπόν της Σλοβενίας. Ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Άλλωστε και πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση γιόρτασε τις πρώτες τις 100 μέρες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι λαμβάνετε τις συστάσεις των Βρυξελών πάρα πολύ σοβαρά και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στην έκθεση του Νοεμβρίου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή περιλαμβάνει και την πρώτη της αξιολόγηση και λέγει ότι η Σλοβενία είναι μία από τις δύο χώρες όπου μία σε βάθος ε, αναθεώρηση θα πρέπει να είναι απαραίτητη. Εγώ νομίζω ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες ξεκάθαρα αποδεικνύουν ότι ξεπεράσαμε τους δείκτες σε δύο τομείς μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταπάντησε βέβαια ότι και αυτό θα πρέπει να προκαλέσει περισσότερο έλεγχο από ό,τι μέχρι τώρα. Πάντως οι μακροοικονομικοί δείκτες και η έλλειψη ισορροπίας είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ σοβαρά. Και θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες απαντήσεις και σε σχέση με αυτά τα οποία υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λεγόμενη Bad Bank. Να θέσω μια επιπλέον ερώτηση στην Σλοβενία πάνω σε αυτό το θέμα το συζητάμε ε, θα έλεγα πάνω από ένα χρόνο και πάνω υπάρχουν νομικά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δημιουργεί και επιπλέον νομικά προβλήματα γύρω από την προσπάθεια αυτή. Τι θα γίνει επιτέλους, έχουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το νομικό πλαίσιο αυτής της τράπεζας ε, που μαζεύει, εν πάση περιπτώσει, ε, τα χρέη των υπολείπων θα λειτουργήσει. ή πιστεύετε ότι απαιτούνται και άλλα μέτρα για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καταρχάς να σχολιάσω λίγο αυτά τα οποία είπατε για τις ανισότητες και την έλλειψη ισορροπίας η Σλοβενία έχει συγκεκριμένες επιδόσεις στον πίνακα αποτελεσμάτων θα έλεγα και έχει δύο τομείς, σε δύο κριτήρια δεν έχει ισορροπήσει τα πράγματα. Μόνο μία χώρα είχε ένα πρόβλημα με ένα αρνητικό αποτέλεσμα και οι υπόλοιπες χώρες είχαν πολύ περισσότερα από δύο αρνητικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά μπαίνει στη διαδικασία περαιτέρω αξιολόγησης. Συμφωνώ ότι στον επιχειρηματικό κόσμο έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και τα προβλήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά η οικονομία πρέπει να ξεπεραστούν γρήγορα. Ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να διαπιστώσουμε αυτά τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, μια πολιτική η οποία να είναι μια πιο μακροπρόθεσμη, βιώσιμη οικονομική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε μια σωστή βάση για να το πετύχουμε. Τώρα για να επανέλθω στο θέμα της λεγόμενης κακής σε εισαγωγικά τράπεζας και το νομικό πλαίσιο. Έχω την αίσθηση ότι τώρα πλέον το νομικό πλαίσιο είναι το ορθό δεν θα μπορούσα να κάνω κάποιο αντίθετο σχόλιο. Αυτό το οποίο είναι υποσυζήτηση όμως τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η ανάγκη να υπάρξει το stress test ε, εκ των προτέρων και η καταγραφή επίσης ε, ε, And doing the test. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει η μεταφορά αυτή ε, πριν γίνουν τα stress test έτσι ώστε να δείξουμε ότι έχουμε προχωρήσει με σωστό τρόπο. Τώρα βέβαια ακούγεται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στα stress test πρώτα και μετά να γίνει η εκαθάριση ουσιαστικά των τραπεζών και η απαλλαγή τους από τις ε, ε, μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε μια κάποια λύση ότι η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και η ποιότητα της σωστής λειτουργίας των τραπεζών είναι κάτι το πιο σημαντικό από την ταχύτητα και αυτό θα προσπαθήσουμε ε, να ε, ικανοποιήσουμε σε μία πρώτη φάση. Σχετικά τώρα με την πιλωτική φάση της μεταφοράς ε, των ενεργητικών των τραπεζών, έχουμε κάνει κάποιες τέτοιες διαδικασίες για να αποδείξουμε ότι οι διαδικασίες οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την κακή σε εισαγωγικά τράπεζα θα λειτουργήσουν κανονικά ή μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά και ότι μπορεί η διαδικασία να γίνει αντικείμενο τακτικής κανονικής διαχείρισης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βολφ Κλίντς από τους Φιλελευθέρους τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσατε να μας δώσετε μια εικόνα κάπως θετική της κατάστασης στη Σλοβενία. Μου φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη θα έλεγα ε, και μερικές φορές ανησυχητική όταν ακούω ότι αρχίζετε να ιδιωτικοποιείτε τις εταιρείες που τώρα είναι κρατικές ακόμα. Αυτό σημαίνει για μένα ότι έχετε χάσει 20 χρόνια. Ε, τα βαλτικά ε, κράτη έπρεπε να αρχίσουν να ιδιωτικοπούν στην αρχή της ανεξαρτησίας τους. Γιατί δεν αρχίσατε ε, νωρίτερα και το γεγονός ότι αρχίζετε τώρα με αργό βήμα, με μικρούς αριθμούς, ε, δεν είναι κάτι το ενθαρρυντικό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, έχουμε την δυνατότητα τώρα να ανακεφαλαιοποιήσουμε ε, τις τράπεζες στην Ευρωζώνη. Έχετε ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ε, μηχανισμό, τον μηχανισμό, τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ή όχι. Και τρίτον, για να βγείτε από τις δυσκολίες σας θα πρέπει να ε, δημιουργήσετε ένα κλίμα το οποίο να είναι ελκυστικό για τους δυνητικούς επενδυτές. Μιλήσατε για τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Θα πρέπει να έχετε διαδικασία λήψης αποφάσεων που να είναι διαφανής, ταχεία, δίκαιη, σωστή, ορθή και να μην έχετε ε, άχρηστη γραφειοκρατία. Εγώ νομίζω ότι έχετε πολλούς υπερβολικά μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό με τρόπο δυναμικό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Λέτε ε, για τα 20 τελευταία χρόνια. Εγώ έχω αναλάβει αυτή τη θέση εδώ και τέσσερις μήνες. Όχι, δεν είναι προσωπική ερώτησή μου. Είναι ερώτηση στον Υπουργό της Σλοβενίας. Ε, την ερώτηση ε, γιατί τώρα και γιατί σε τόσο μικρούς αριθμούς όταν βλέπουμε την ιδιωτικοποίηση πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή με ρεαλιστικό τρόπο, πραγματιστικό τρόπο. Υπήρξαν ε, προσπάθειες πολιτικοποίησης ε, στην Σλοβενία πάρα πολύ συχνά και συζητήθηκαν τα θέματα αυτά ε, και η έναρξη της αυτής της διαδικασίας. Έγινε σε πολύ μικρούς αριθμούς, σε πολύ περιορισμένη έκταση. Είχαμε την επιλογή να αρχίσουμε μια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση και να έχουμε όλον τον κατάλογο των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αποκρατικοποιηθούν, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει αμέσως στην αγορά. Δεύτερο, μπορούσαμε να αρχίσουμε μια μακρά ε, συζήτηση που, που χρειαζόταν ένα ε, πολύ χρόνο για να καταλήξει σε μια απόφαση. Έχουμε έναν κατάλογο πέντε εταιριών και ο, κα, ο κατάλογος ε, έγινε 15. Ε, εμείς καταρτίζουμε τον κατάλογο ούτως ώστε να, έχει, ε, να είναι ορθολογιστικός να πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτόν τον κατάλογο και να δούμε ε, τι είναι εφικτό σε αυτό τον τομέα και θα πρέπει επίσης να έχουμε έναν ταχύ ρυθμό, να αρχίσουμε αμέσω, αλλά όταν αρχίζει η διαδικασία, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να μεγιστοποιεί την αξία των επιχειρήσεων αυτών προς όφελος των φορολογουμένων θα πρέπει να πουληθούν οι εταιρείε αυτές ώστε να μεγιστοποιηθεί το εισόδημα. Αυτή είναι η εξήγηση. Επίσης συμφωνήσαμε και υποσχέθηκα στο Σλοβενικό Κοινοβούλιο ότι θα προετοιμάσουμε όλη την στρατηγική με όλο τον κατάλογο των επιχειρήσεων που προσδιορίζονται ως εταιρείε προς ιδιωτικοποίηση και ότι θα έχουμε μια συζήτηση για την στρατηγική, για το τι εταιρείε είναι στρατηγική σημασία ούτως ώστε να παραμείνουν κρατικές και τι, ποιες είναι καλύτερα να ιδιωτικοποιηθούν. Προγραμματίζουμε μια τέτοια συζήτηση στο φθινόπωρο. Ε, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δεν χρησιμοποίησαμε τις διευκολύνσεις αυτές. Θελήσαμε να κάνουμε με δικά μας μέσα, με τα ίδια μέσα, να ανακεφαλαιοποιήσουμε. ούτω ώστε να κάνουμε αυτήν τη διαδικασία, να προβούμε σε αυτή τη διαδικασία ε, μόνοι μας, ε, διότι καλύτερα και απέναντι στους εταίρους μας, να μην χρησιμοποιήσουμε τα δικά τους κονδύλια για δικούς μας σκοπούς. Σχετικά για το κλίμα, για δυνητικούς επενδυτέ, νομίζω ότι η ιδιωτικοποίηση είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το άνοιγμα αυτό. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει στο παρελθόν που δεν είναι πολύ ορατά ε, το κλίμα στην Σλοβενία από την άποψη της ε, δίκησης δεν είναι πολύ προβληματική εικόνα, βέβαια πάντοτε μπορεί να βελτιωθεί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Για μένα έχουμε δύο προτεραιότητες πρώτα ε, και σε αυτές εστιάζομαι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η ερώτησή μου, ε, μάλλον δύο ή τρεις ερωτήσεις, είναι πάρα πολύ απλές. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Σλοβενία είναι μια από τα 11 μέλη που κάνουν την πρόταση σχετικά με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με ενισχυμένη, για συνισχυμένη συνεργασία. Και αυτή είναι το πρώτο ερώτημά μου. Ποιο είναι το μέγεθος της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Σλοβενία. Δεύτερη ερώτηση, ποια είναι τα αναμενόμενα έσοδα που αναμένεται να εισπράτεται από τον φόρο αυτό. Και η τρίτη ερώτηση, διότι μιλάτε για δυσκολίες και εγώ εκτιμώ, πράγματι εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο η Σλοβενία θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο εσωτερικό της Σλοβενίας. Πού θα προτιμούσατε να διοχετεύσετε τα έσοδα που θα προέλθουν από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στον προϋπολογισμό της Σλοβενίας ή στον προϋπολογισμό τον Ευρωπαϊκό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση θα έχω τον ακριβή αριθμό της αγοράς της Σλοβενικής. Δεν έχω τα στοιχεία αυτά μαζί μου. Ε, η αγορά είναι αρκετά μικρή και δεν νομίζω ότι θα έχουμε τεράστια έσοδα από αυτό το φόρο. Βεβαίως ε, δεν βασιζόμαστε σε αυτά τα έσοδα, σε αυτό το εισόδημα ε, στο, για τα δημόσια οικονομικά μας, διότι είναι κάτι το αβέβαιο. Έχουμε μια άλλη παρόμοια, έναν άλλο παρόμοιο φόρο για τις τραπεζικές υπηρεσίες που εισήχθη ε, πέρυσι, αλλά και το εισόδημα από το φόρο αυτό δεν είναι σημαντικό. Δεν βασιζόμαστε λοιπόν ακόμη σε αυτά τα έσοδα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα αποφασίσουμε πού θα διοχετευτούν αυτά τα χρήματα, για πού θα προορίζονται. Ε, δεν έχω ακόμα τα σχετικά στοιχεία, θα τα έχω αργότερα. Από τους πρασίνους τώρα, ο Φιλίπ, εσύ ή ο Σβέν. Ο κύριος Γκίγκολτ, εγώ είμαι πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθατε Υπουργέ. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας το εξής, διότι δεν υπόθηκε ακόμα. Νομίζω ότι η Σλοβενία είναι μια χώρα που όχι μόνο είναι όμορφη, αλλά και από οικονομική προοπτική είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι καταφέρατε μετά την πτώση του σιδηρού ε, παραπετάσματος, καταφέρατε εσείς να βγείτε από αυτή τη δύσκολη περίοδο πολύ πιο αλόβητη από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το κατακεφαλήνα έψαση υψηλότερο δεν επαναλάβατε πολλά από τα σφάλματα που έγιναν αλλού. Your human development index is... Και η ε, ανάπτυξή σας η ανθρώπινη ε, γενικότερα είναι πολύ πιο ψηλή από άλλες χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ε, μπορείτε να είστε περήφανοι γι' αυτό και θα πρέπει να το πούμε κι εμείς. Και να είμαστε και λίγο προσωπικοί, προσεκτικοί, συγγνώμη, λέγοντας γιατί δεν κάνατε πιο γρήγορα ιδιωτικοποιήσεις κτλ είναι ένας από τους λόγους, γιατί ακριβώς ήταν πιο επιφυλακτική και πιο συγκρατημένη η πολιτική. Και γι' αυτό η Σλοβενία ε, ήταν ε, διαφορετική και ήταν και η ζωή των πολιτών η καθημερινή πολύ καλύτερη από που αλλού. Αλλά νομίζω ότι παραχαρώσατε όμως τελικά ε, και δεν καταβάλατε πολύ μεγάλες προσπάθειες στη συνέχεια. Έρχομαι τώρα στις λιγότερο ευγενικές ερωτήσεις. Ε, πρώτον, μεταρρύθμιση ε, του συνταξιοδοτικού συστήματος. Έχετε ένα πρόβλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία, κάνατε μεταρρυθμίσεις, αλλά τι θα γίνει για την περίοδο μετά το 2020. Μιλήσατε και για το κομματικό σας σύστημα και την ιδιαίτερη λειτουργία του πολιτικού συστήματος ε, και την έκφραση. Και επίσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είστε εκτός στόχων. Το ποσοστό της συμμετοχής των ανανεώσιμων στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ε, δεν είναι στα πλαίσια των στόχων και πώς θα δρέψετε καρπούς εσείς από τα πλεονεκτήματα της πράσινης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Να αρχίσω από τη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος. Πέρυσι έγινε αυτή. Έφερε κάποια αποτελέσματα. Μερικά όμως. Όχι συνολικά. Το ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας ε, δρόμο. Το έχω υπόψη μου. Αλλά θα πρέπει πρώτα να σταθεροποιήσουμε τις οικονομικές μας δραστηριότητε και μετά. Διότι εξήγησα αυτή τη δομή των τριών πυλώνων και πώς θέλουμε να λαμβάνουμε τις οικονομικές αποφάσεις το βραχυπρόθεσμο και την αναδιάρθρωση αργότερα μέσω μακροπρόθεσμη. Να κάνω μια σύγκριση ε, με ένα αεροπλάνο. Πρώτον πρέπει να αποφασίσεις ποιος θα είναι ο κυβερνήτης. Μετά να σταθεροποιήσεις το ύψος το οποίο πετάς. Και το τρίτο είναι η κατεύθυνση προς τα που θες να κατευθυνθείς. Ε, ε, το πρώτο λοιπόν είμαστε τώρα στην σταθεροποίηση του ύψους και στο ποιος θα είναι ο πιλότος. Ε, και με ποιο τρόπο θα κυβερνήσει το αεροσκάφος. Μετά θα πάμε στην κατεύθυνση. Το θέμα λοιπόν της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ε, είναι στο τρίτο πυλώνα. Δεν είναι πάρα πολύ ε, άμεσο και αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον να προέχει η σταθεροποίηση. Δεύτερη ερώτηση για το κομματικό σύστημα. Είναι στο δεύτερο πυλώνα. δεν τα έχουμε λύσει όλα. Εργαζόμαστε ακόμα για την διοίκηση επιχειρήσεων και τη διακυβέρνηση, αλλά το κομματικό σύστημα θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, πώς ε, θα ανεβάσουμε το κατόφλι για να μπαίνουν λιγότερα κόμματα στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση κατ' επέκταση. Η πολιτική σταθερότητα ε, θα πρέπει επίσης να είναι κάτι δεδομένο και μόνιμο στη Σλοβενία. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να εργαζόμαστε προς τα εκεί. Ούτε είναι θέμα του Υπουργού Οικονομικών. Ε, αυτό ελπίζω να καταλήξω. Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες ενέργειες, τι κάνουμε αυτό τον καιρό. Θέτουμε στόχους και προτεραιότητες. Τι περικοπές θα κάνουμε στον προϋπολογισμό και πού. Και δυστυχώς έχουμε περικόψει πάρα πολλές επενδύσεις και δι επενδύσεις σε ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας επίσης. Εδώ είναι μια ελαφρά, ε, ε, ε, λεπτή ισορροπία. Από τη μια θα πρέπει να ισορροπιστεί, να ισοσκελιστεί ο προπολογισμό και από την άλλη να δούμε και τα διορθωτικά. Να τηρήσουμε την πειθαρχία και τη χρονική. ο Γιώργιον Κλούτε από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη και την προθυμία να κάνουμε διάλογο εδώ. Μισό λεπτό να βάλει τα ακουστικά σας, ναι, γιατί μιλάω γερμανικά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και για την προθυμία να συζητήσετε μαζί μας. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη προς την Προεδρία του Συμβουλίου του Λιθουανία. Αυτό τον καιρό έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό και τη διαφάνεια ως προς τα τραπεζικά τέλη. Είναι μικρό μεν το θέμα, το ξέρω ότι δεν κυριαρχεί, παρόλα αυτά ε, είναι σημαντικό πριν τα τέλη της θητείας να εγκριθεί και στον τριμερή διάλογο. Εμείς απευθυνθήκαμε στην Προεδρία ως συντονιστές με την παράκληση να μπει ή δυνατόν στον κατάλογο προτεραιοτήτων και θέλω να ρωτήσω εσάς εσείς πώς φαντάζεστε ε, μπορέσουμε να το συζητήσουμε, θα προλάβουμε στην παρούσα θητεία. Και ένα δεύτερο γενικότερο ζήτημα για την οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που είναι σε κρίση τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες ε, όλο και περισσότερο συζητούμε για τα προγράμματα ε, των περικοπών και των εξοικονομήσεων. Δεν αρκούν οι περικοπές, χρειάζεται και ανάπτυξη εκτός από τη λιτότητα. Ε, εσείς πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει και μπορεί να τονωθεί η ανάπτυξη στις χώρες μέρες, ε, ιδιαίτερα στις χώρες που περνούν κρίση, γιατί μόνο η εξοικονόμηση δεν αρκεί για να ξεπεραστεί η κρίση και η ανάπτυξη είναι πραγματικά ένα ουσιαστικό στοιχείο εδώ. Μέχρι τώρα έχω την εντύπωση ότι στο Συμβούλιο το στοιχείο αυτό της ανάπτυξης δεν κυριαρχεί πάρα πολύ όσο εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Uh, thank you for the two uh, Σας ευχαριστώ για τις δύο ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, το πρώτο αφορά τη διαφάνεια για τους τρόπους αλλαγής λογαριασμών και τη διαφάνεια των τραπεζών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε υπό εξέταση στη Σλοβενία. Και το δεύτερο είναι το πώς θα περάσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης εμείς οι χώρες που έχουν δυσκολίες. Για το πώς μπορεί να αλλάξει κανείς τράπεζα και λογαριασμό και διαφάνεια των λογαριασμών. Υπήρξε κάποια δράση στη Σλοβενία για το θέμα αυτό από την Κεντρική Τράπεζα για να διευκολυνθούν οι πελάτες να αλλάζουν τράπεζα. Και νομίζω ότι έχουν ένα απλό τρόπο για να το κάνουν αυτό. Μπορούν να περνούν από τη μία τράπεζα στην άλλη. Αυτό είναι κάτι που έχει λοιπόν γίνει. και δεν νομίζω ότι είναι ένα από τα κομβικά θέματα που έχουμε μπροστά μας τώρα. Το δεύτερο, τι εναλλακτικέ υπάρχουν στη δημοσιονομική λιτότητα για να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό που έχει σημασία, και μιλάω για τη δική μου χώρα, η Σλοβενία είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία, η ανταγωνιστικότητά της είναι σημαντική. αν δω το σύνολο της Ευρωζώνης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη οικονομική περιφέρεια. Στη Σλοβενία το 60 με 80% των καταναλωτικών προϊόντων εισάγεται και το 60% εξάγεται. Η δημοσιονομική λιτότητα λοιπόν είναι λογική εφόσον καλύπτει τις δαπάνες, όταν μειώνει το κόστος, καθιστά στη χώρα πιο ανταγωνιστική. Και νομίζω ότι το σύνολο της περιφέρειας ε, θέλει να υπάρξει λιγότερο λιτότητα, αν θέλετε, αλλά σε επίπεδο περιφερειακό, σε επίπεδο μιας μικρής οικονομίας κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Το θέμα είναι να προσπαθήσει να συνδυάσει κανείς τα διάφορα οικονομικά στάδια και τις οικονομικές πολιτικές. Η τρέχουσα κατάσταση λέει ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα του τραπεζικού τομέα, ε, προς το παρόν τα επιτόκια και σε σχέση για τις καταθέσεις και σε σχέση με τα δάνεια είναι πάρα πολύ ψηλά παρά τις περιοριστικές ε, ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και απ' την άλλη πιέζουμε και δημοσιονομικά. Αυτά τα δύο καθιστούν την ανάπτυξη δύσκολη. Θα πρέπει να μπορέσει κανείς να είναι χαλαρός σε σχέση με την νομισματική πολιτική, να ξεκαθαρίσει το ισοζύγιο, να χαμηλώσει το πραγματικό κόστος, να είναι ρευστή η οικονομική δραστηριότητα, να υπάρχει δυνατότητα πίστοσης και μετά να περάσει κανείς τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ο χρονισμός με λίγα λόγια των οικονομικών πολιτικών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν λαμβάνονται, ε, όταν εξετάζονται οι περιφερειακές χώρες. Προσπαθούμε εμείς να ξεκαθαρίσουμε τις τράπεζες σε μια πρώτη φάση για να μπορέσουμε να περάσουμε εκ των υστέρων στη δημοσιονομική πειθαρχία. Ευχαριστώ. Πέτερ λέει. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε ε, και για την παρουσίασή σας και για την παρουσία σας. Ξέρετε τι πιστεύω εγώ για τη τραπεζική κρίση. Βρισκόμαστε σε μια κρίση γιατί ήταν ε, η πολιτική που κυριαρχούσε στο τραπεζικό σύστημα. Δεν παίζαμε ούτε με τους αγώνες της αγοράς, ούτε της χρηματαγοράς, ούτε του συμφέροντος του κρατικού. Δίνανε δάνεια, θαλασσοδάνεια, χωρίς καμία εγγύηση. Τι σπταίει τώρα. Όχι αυτοί που πληρώνουν την κρίση. Επίση, τι θα γίνει με το πράσινο φω για τι μεταφορές πιστώσεων. Επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει, αλλά τα πράγματα διαφέρουν στις Βρυξέλλες σε σχέση με τη Λιουμπλιάνα ή οι δηλώσεις. Η Λιουμπλιάνα λέγει ότι ε, θα γίνουν γρήγορα οι δηλώσει. Ε, των πιστώσεων αυτών. Ε, οι Βρυξέλλες λέγουν ότι θα πρέπει πρώτα να καθαρίσουν οι λογαριασμοί. Τι έγινε, έχετε συμφωνήσει Λιουμπλιάνα και Βρυξέλλες για το τι πρέπει να γίνει για τη διαφάνεια και ποιος περιμένει ποιον. Τηρείτε μια στάση αναμονής εκεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Νομίζω ότι στις δύο προηγούμενες απαντήσεις μου ε, απάντησα, κάλυψα εν μέρη τα όσα ρωτήσατε. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Κοιτάξτε, όλα αυτά που κάνουμε εμείς για να στήσουμε αυτή την Bad Bank, την τράπεζα των επισφαλιών, ε, είναι σε γερά θεμέλια. Εξασφαλίζουμε σωστές διαδικασίες. Ε, έτσι, ακριβώς ώστε να ε, προστατεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων. Θέλουμε η διαδικασία να είναι πάρα πολύ σαφής, πάρα πολύ διαφανής και όσο γίνεται να ε, ε, αξιοποιήσουμε τη διεθνή εμπειρία. Και μάλιστα με πάρα πολύ ε, γρήγορες διαδικασίες, γιατί και ο χρόνος είναι χρήμα, ως γνωστόν. Η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων δεν έχει να κάνει μόνο με τη μεταφορά αυτή των πιστώσεων. Θα πρέπει να γίνουν γρήγορα διαδικασίες για να μην χάσουμε ευκαιρίες. Ε, και να μην χάσουμε και μελλοντικές ευκαιρίες για να επανέλθει η ανάπτυξη. Λοιπόν, ε, όλη η διαδικασία ακριβώς είναι αφιερωμένη σε αυτό και αφοσιωμένη στην προστασία των ε, χρημάτων των φορολογουμένων. Τι γίνεται με τη μεταφορά των ποσών και το χρονισμό. Βεβαίω θέλουμε πολύ γρήγορα να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του θέρου, το είπα και προηγουμένως άρρωστε, Σχεδιάζαμε η πρώτη δόση να έρθει πριν τα τέλη Ιουνίου ε, ήταν η πιο εύκολη διαδικασία για τη φερεγγιότητα, αλλά όταν συζητήσαμε τις συστάσεις αναχώρα, αποφασίσαμε να κάνουμε πρώτα τα τεστ τεστ και την αθεώρηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και πρόσφατα συμφωνήσαμε ότι είναι καλύτερο να μην ε, προχωρήσουμε σε βεβαιασμένες κινήσεις. και όχι οπωσδήποτε να έρθει πρώτη δόση το καλοκαίρι, αλλά να αναθεωρήσουμε πρώτα, να εκτιμήσουμε τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών, να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να κάνουμε τα stress test και την πιλωτική μεταφορά για να εξασφαλιστεί η σωστή διαδικασία στο σύνολό της Και νομίζω αυτός είναι ο σωστός ε, τρόπος ε, να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Κυρία Κλέβα. Yes. Yes. Ναι. Ε, πιστεύω ότι ο υπουργό ε, δεν μπορεί να απαντήσει για τα 20 τελευταία χρόνια, για αυτό που έχει γίνει τα 20 τελευταία χρόνια, αλλά μπορώ να τον ρωτήσω για τα σημερινά θέματα, τα επίκαιρα, τα οποία ακόμη δεν συζητήσαμε. Θα ήθελα να μιλήσω για την κερδοσκοπία και τις ε, υποθέσεις που γίνονται για τη Σλοβενία με την κατάρρευση της Κύπρου. Πρέπει να αντιδράσουμε, να αντιδράσουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε σε αυτήν την Επιτροπή δεν είμαι ε, πολύ υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων και νομίζω ότι ο κατάλογος των 15 επιχειρήσεων που ε, θα προταθούν για ιδιωτικοποίηση αυτό έγινε κάπως βεβιασμένα πολύ γρήγορα. Δεν νομίζω ότι έχει ε, υπάρξει επαρκής σκέψη ε, σχετικά με αυτόν τον κατάλογο. Μια άλλη ερώτηση είναι η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που αναφέρατε εσείς και που ανέφεραν και συνάδελφοί μου. Σχετικά με την ανεργία των νέων είμαι ε, σοσιαλδημοκράτησα και νομίζω ότι δεν κάναμε τίποτα τίποτα για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Νομίζω ότι στην επόμενη μεταρρύθμιση και θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό η Σλοβενία. Μια ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση η ανεργία των νέων. Uh, Uh, uh, Σχετικά με την αγορά εργασίας και την ανεργία των νέων, το καλύτερο uh, που να κάνουμε είναι να επανέλθουμε στην ανάπτυξη, διότι η ανάπτυξη είναι για όλους, όχι μόνο για τους ενήλικες, τους μεγάλους, αλλά και για τους νέους να έχουμε καλύτερο ισολογισμό των τραπεζών, να αναδιαρθρώσουμε ε, και να εξηγιάνουμε τα δημοσιονομικά μας. Ήταν η τελευταία ερώτηση. Θέλετε τίποτα άλλο να προσθέσετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι πάντα δύσκολο να έρχεστε, νομίζω, έτσι στο τέλος του απογεύματος, αλλά δεν είναι το τέλος, διότι θα έρθει και ο Υπουργός Οικονομικών της Λιθουανικής Προεδρίας. Θα έχουμε τώρα μια, ένα διάλειμμα δύο-τριών λεπτών και μετά θα επανέλθουμε.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 Πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που καλωσορίζω τον Υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας εδώ στην συνηθισμένη ανταλλαγή απόψεων στην αρχή της κάθε Προεδρίας ούτως ώστε να ασχοληθούμε με θέματα που σχετίζονται με τις προτεραιότητες όπως όλοι γνωρίζουμε η Προεδρία γνωρίζει πολλά περισσότερα για τους φακέλους στο τέλος της Προεδρίας από ό,τι στην αρχή, αλλά περιμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας και την παρουσία σας. Θα έχετε 10 λεπτά και μετά θα έχουμε την συνήθη συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας δώσω όμως το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα, σύμφωνα με την καλή ευρωπαϊκή παράδοση, να αρχίσω στα λιθουανικά, στην ματρική μου γλώσσα που είναι από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας ζητώ λοιπόν να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σας ευγνωμονώ πολύ για την ευκαιρία που δίδετε ε, να σας ε, παρουσιάσω σήμερα τη Λιθουανική Προεδρία για τα θέματα ε, οικονομικών και δημοσιονομικών. Επιτροπή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ε, από νομοθετικής πλευράς και ιδιαίτερα για το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στο οποίο θα προεδρεύσω το επόμενο εξάμεινο. Και προσβλέπω και ελπίζω σε μια επικοδομητική συνεργασία ευθύ εξ αρχής από την αρχή της Προεδρίας μας. Προφανώς, πριν πω στις προτεραιότητες ε, της ε, Προεδρίας, οφείλω να ε, ευχαριστήσω την Ιρλανδία. Το πρώτο μέλος του τρίου της Προεδρίας ε, για ε, την εξαιρετική εργασία τους. Και βλέπω και από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πόσο ήταν το έργο της Προεδρίας. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο περίμενε περισσότερα αποτελέσματα από την Ελλανδική Προεδρία αλλά δεν θα πρέπει καθόλου να υποτιμούμε ε, τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα ζητήματα και σημαντικά. Ε, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που έχουν μπει τώρα πλέον γερά θεμέλια για τη δική μας Προεδρία για να συνεχίσουμε την προσπάθεια της Ιρλανδικής. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία ε, θα συζητηθούν στον τριμερή διάλογο και μπορούν να αρχίσουν και να συνεχίσουν οι εντατικές ε, συνομιλίες ήδη από τον Ιούλιο. Προεδρεύοντας το ΕΚΟΦΗΝ θα κάνω ό,τι μπορώ και θα φροντίσω πάντα να ε, πριτανεύει η συνένεση, το επικοδομητικό πνεύμα, να έχουμε αποτελεσματική δράση και ελπίζω και η ομάδα μου να είναι πάρα πολύ και αρκετά φιλόδοξη. γιατί έχει και αυτό τη σημασία του για όλους μας και στο Κοινοβούλιο και στις πρωτεύουσε και παντού για τους πολίτες της Ευρώπης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή όλους ιδιαίτερους. Η αποτελεσματική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προσωπική μου προτεραιότητα. Προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη για την αποτελεσματική συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ μεγάλες οι οικονομικές προκλήσεις. Η εξηγίαση των προϋπολογισμών, ε, ο ισοσκελισμός τους είναι πάρα πολύ σημαντικός για να υπάρχει ε, βιώσιμη οικονομία. Θα πρέπει να επανακτήσουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και να ενισχύσουμε και την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα. Αλλά βασικός στόχος για όλους μας θα πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη. Το επόμενο εξάμεινο Θα πρέπει να εμφανιστεί ήδη η ανάπτυξη. Έχουν ληφθεί οι πρώτες σημαντικές αποφάσεις και έχει έρθει η ώρα των αποτελεσμάτων. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να χαρώσουμε τις προσπάθειές μας ή ε, την προσοχή μας. Παραμένουμε ε, σε παγρύπνηση για να υλοποιηθούν αυτές ε, οι προγνώσεις για να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορούν να δημιουργούνται ξανά θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους. για να μπορούν οι πολίτες να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Συνεχίζω στα αγγλικά. Η Προεδρία μας βασίζεται στα θέματα που θα εξασφαλίσουν αξιόπιστη, αναπτυσσόμενη ε, και ανοιχτή Ευρώπη. Βεβαίως ε, η ΕΚΟΦΗΝ ασχολείται με πολλές από αυτές τις προτεραιότητες διότι ε, για μένα η βασική προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη στην Ευρώπη αλλά αξιοπιστία είναι αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε υιοθετώντα κατάλληλες νομοθετικές πράξεις και αυτά θα είναι πραγματικά μέσα τα οποία θα έχουμε στα χέρια μας. Σήμερα υπήρξαν ε, δύο πολύ εντυπωσιακά γεγονότα. Κατά τη διάρκεια του ΕΚΟΦΗΝ μπόρεσα να καλωσορίσω την Κροατία ως νέο μέλος της οικογένειάς μας, το 28ο μέλος της οικογένειάς μας και πριν από μία ώρα συμμετείχα στην, στους εορτισμούς, σήμερα στην ΕΚΟΦΗΝ υιοθετήσαμε ε, νομοθετικές πράξεις ε, τρία, ε, τρίας κανονισμούς για την προσχώρηση της Λετωνίας στην Ευρωζώνη. Όλε μπορώ και εγώ να χειροκροτήσω διότι ήταν για μένα προσωπικά σημαντικό. Είναι τιμή, είναι προνόμιο αλλά είναι και μεγάλη χαρά για μένα και είναι επίσης μια πρόκληση για τη Λιθουανία. Έχουμε ενώπιόν μας τον ορίζοντα του 2015 για να υιοθετήσουμε το ευρώ. Θέλει να είμαστε οι επόμενοι. Ζηλεύουμε κάπως βλέποντας τη Λετωνία. Εδώ, αν μου το επιτρέπετε, θα ήθελα να ζητήσω και τη δική σας ε, υποστήριξη σε αυτό το εγχείρημά μας, σε αυτή την προσπάθεια, διότι αυτό ε, δεν, δεν είναι μόνο συμβολικό, αλλά είναι κάτι το πρακτικά σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται, επεκτείνεται, η Ευρωζώνη επίσης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η Ευρωζώνη ε, και το εγχείρημα της Ενωμένης ΕΕ είναι κάτι το αξιόπιστο. Οι λαοί πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ιδέα. Οι χώρες πιστεύουν στο ευρώ ως κοινό νόμισμα. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, θεμελιώδες εγχείρημα βαρύνουσας σημασίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτές τις ιδέες όταν μιλάμε για τις τεχνικές λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές, αλλά οι βασικές ιδέες θα πρέπει ε, πάντοτε να τις ακολουθούμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και υγιή δημόσια οικονομικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα ήθελα να συγκεντρωθώ σε μερικούς από τους φακέλους που για μας θεωρούνται σημαντικοί σε συνεργασία μαζί σας, διότι εσείς είσαστε συνομοθέτες σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες. Γι' αυτό περιμένω αφού μίλησα, συνομίλησα με πολλούς από εσά πριν από την Προεδρία μας, πολλούς από εσά μέλη ε, της Επιτροπής ΕΚΟΝΟ ότι τα θέματα αυτά είναι εξίσου σημαντικά για σας. Νομίζω, βεβαίως, πρέπει να κάνουμε πρόοδο ε, σημαντική ε, σε πάρα πολλές νομοθετικές προτάσεις ευρύτατες κυρίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κυρίως σε σύνδεση με την Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι η, ευρωπα ε, η... Τραπεζική Ένωση και τα δημοσιονομικά και η οδηγία κυρίως ανάκαμψης και εξυγίασης των τραπεζών που αύριο θα συζητηθεί σε τριμερή διάλογο, ήδη αύριο, αφού θα έχουμε επιτύχει ένα δύσκολο συμβιβασμό στο ΕΚΟΦΗΝ, νομίζω όμως ήταν δίκαιο συμβιβασμό τώρα έχουμε αυτό το φάκελο που πρέπει το θέμα αυτό να προωθήσουμε. Επίσης έχουμε το σύστημα εγγύησης εξασφάλισης των καταθέσεων. Προτιθέμεθα να προωθήσουμε τα δύο θέματα αυτά μαζί παράλληλα. Και βεβαίως ο μηχανισμός, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός μπορώ να σας ενημερώσω ότι σήμερα η Επιτροπή μας διαβεβαίωσε ότι η πρόταση για ε, τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης ε, θα παρουσιαστεί αύριο η πρόταση. Η Επιτροπή βεβαίως και αυτή πρέπει να προχωρήσει. Ενώνοντας ε, τις προσπάθειές μας νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτού του πολιτικού κύκλου, δηλαδή μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές. Η οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι μέτρα ριζικά έχουν πρόσφατα υιοθετηθεί υπό τη μορφή του, της νομοθεσίας και 2 pac το, ε, Συμβούλιο των Υπουργών που προεδρεύω είναι ευγνώμων για τον συμβιβασμό που επιτεύχθη στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα ε, θα πρέπει να δράσουμε, ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως τα νομοθετήματα αυτά. Και συμφωνήσαμε σήμερα μερικά νομικές πράξεις που θα εξασφαλίσουν την συνεργασία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου του, για την εξάντε αξιολόγηση των ε, προϋπολογισμών των κρατών μελών και βεβαίως ε, έχουμε επίσης ε, τις ειδικές συστάσεις αναχώρα και όλα τα περίπλοκα μέτρα που συνδυάζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα αποδώσουμε την πρέπουσα προσοχή όχι μόνο για ε, την ε, εφαρμογή αυτών ε, των διαδικασιών. Θα εξετάσουμε ενδελεχώς και θα επανέλθουμε στο ΕΚΟΦΗΝ για αξιολόγηση των παρουσών διαδικασιών για να αξιολογήσουμε εάν είναι οι κατάλληλες, είναι αποτελεσματικές ή όχι, αν αποδίδουν αποτελέσματα ή όχι, αν είναι απλή γραφειοκρατία ή αν είναι πράγματι κάτι με οικονομικό νόημα για τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή να είναι μια εμπειρία πάρα πολύ χρήσιμη για το ΕΚΟΦΗΝΑ και ε, είμαι αποφασισμένος ε, να μοιραστώ αυτήν την εμπειρία με τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας. Το μέσο του ισοζυγίου πληρωμών θα το αναφέρω ε, για τα κράτη-μέλη που δεν είναι στην Ευρωζώνη σύμφωνα με την νομοθεσία του ΠΑΚ νομίζω ότι είναι από τις προτεραιότητες μας, ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Πρόκειται για έναν σημαντικό μηχανισμό, όχι μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά και για αυτούς που είναι εκτός. Πρέπει να εργαστούμε για την Ευρώπη των 28 και αυτό είναι μια άλλη από τις ισχυρές μου προτεραιότητες. Είναι ουσιαστικό η ευρωπαϊκή οικονομία να επωφεληθεί από υγιείς αγορές ανθεκτικές και διαφανές που εργάζονται προς το συμφέρον των φορολογουμένων. Είμαστε όλοι ε, φορολογούμενοι, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί και η προστασία των επενδυτών, πράγμα που είναι σημαντικό για την οικονομία. Ε, γι' αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στην οδηγία MIFID για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως επίσης ε, και για τον κανονισμό των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και έχουμε στους τριμερείς διαλόγους θα προωθήσουμε αυτούς τους φακέλους που έχουν υψηλή προτεραιότητα. Μπορώ να σας πω ότι είναι ήδη εφικτό να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, για τον φάκελο Omnibus 2 που είναι σημαντικό για την ασφαλιστική αγορά τώρα που η Κομισιό έχει εκδώσει την έκθεση για την ε, τεχνική αξιολόγηση από την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή για τις ασφάλειες και τις επαγγελματικές συντάξεις μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από την ενία αγορά θα κάνουμε μπορούμε για να προωθήσουμε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, για έναν απλό λόγο, διότι είναι μια οδηγία για τους καταναλωτές. Και νομίζω ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον όλων μας να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες που θα θεωρηθούν αμέσως επωφελείς από τους πολίτες. Τώρα θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για την φορολογία όπου έχουμε το πρόβλημα να έχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο, αλλά όπου είμαι απόλυτα βέβαιος και θα σας ζητήσω την υποστήριξή σας. Πρέπει να έχουμε την ισχυρή πολιτική σας υποστήριξη κατά πολέμηση της φοροδιακατά της διαφυγής και της φορολογικής απάτης είναι ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων και διεθνώς νομίζω στην ατζέντα διεθνώς έχει ψηλή προτεραιότητα. Έχουμε ήδη ε, ε, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε ευγνώμονες για τα ψηφίσματα αυτά διότι ήσασταν απόλυτα σαφείς για το θέμα και νομίζω ότι όλοι κατανοούν ότι πρόκειται για ε, μια πραγματική προτεραιότητα να εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα τα οποία είναι κλεμμένα, να εξασφαλίσουμε ότι όλοι πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο ε, φόρων, ακόμα και οι πολυεθνικές εταιρείες. Φιλόδοξο σχέδιο για την αυτόματη ανταλλαγή ε, τραπεζικών πληροφοριών και αυτό περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την οδηγία αποταμιεύσεων και επίσης την οδηγία διοικητικής συνεργασίας που βρίσκονται τώρα επιτάπητος. Είναι σημαντικές πρωτοβουλίες και θα ζητούσα τα μέλη της Επιτροπής να μας υποστηρίξουν πολιτικά σε αυτό το τομέα. Έχουμε επίσης και άλλους φακέλους φορολογικούς Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Θα κλείσω πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διαταξή μας πρόκειται για τον προϋπολογισμό τον Ευρωπαϊκό 2014. Είναι έργο μιας άλλης επιτροπής, αλλά είναι και αρμοδιότητα ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι για τους γραφειοκράτες, δεν ε, είναι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί. Κάνουμε κάτι για το λαό, αν δεν έχουμε τον κατάλληλο προϋπολογισμό την 1η Ιανουαρίου αυτό μπορεί να σημάνει ότι πάρα πολλά σχέδια και προγράμματα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν θα χρηματοδοτηθούν καταλήλως. Είναι προτεραιότητα για μας. Θα, δεν θα αφιστούμε καμιάς προσπάθειας ούτω ώστε να έχουμε συμβιβασμούς και συμφωνία με στα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως είναι επίσης ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου και από ό,τι καταλαβαίνω τακτικές ανταλλαγές απόψεων με εκπροσώπους εθνικών κυβερνήσεων επίσης ε, και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπονται και είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι μια άλλη δυνατότητα το τρίτο ευρωπαϊκό εξάμεινο τελείωσε με τις ειδικέ συστάσεις που σήμερα υιοθέτησε το Συμβούλιο για τις χώρες. Βεβαίως είναι σημαντικό βήμα, βεβαίως έχετε πολλές ερωτήσεις και εγώ έχω πολλές ερωτήσεις για πώς, το πώς αυτές οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα θα υλοποιηθούν. Συμφωνώ με τις κριτικές ότι καμιά φορά δεν είναι πολύ συγκεκριμένες, αλλά νομίζω ότι είναι το τρίτο ευρωπαϊκό εξάμεινο και ότι το τρίτο ήταν καλύτερο από το δεύτερο. Νομίζω ότι το τέταρτο ευρωπαϊκό εξάμεινο που θα αρχίσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας θα είναι πολύ πιο οργανωμένο, πολύ πιο ουσιαστικό και ότι θα επιφέρει ορισμένες καινοτομίες. Επίσης, λόγω του Τούπακ και ε, Περιμένω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία μαζί για τα θέματα αυτά. Είναι μεγάλη λοιπόν τιμή και ευθύνη για τη χώρα μου. Η πρώτη από τις βαλτικές χώρες που ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου και αισθάνομαι πράγματι κάπως φοβισμένος Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής περίοδου, γι' αυτό συνάντησα πολλούς τους, από τους συναδέλφους ε, μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκονται εδώ και σας ζητώ περαιτέρω συνεργασία. Ε, προσωπικά εγώ αισθάνομαι ότι είναι προσωπική μου ευθύνη να εξασφαλίσω μια αγαστή συνεργασία μαζί σας Καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε ε, στη Λιθουανία τον σημαντικό, τον σημαντικότατο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ε, μπορεί ε, να συγκεράσει τις διάφορες θέσεις για να έχουμε μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή ιδέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που ξεπέρασα τον χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Και τώρα ε, περιμένω τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένουμε να υπάρξει συνεργασία μαζί σας. Εδώ και πέντε χρόνια από τότε που, ε, που πέρασε η έκθεσή μου για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών σε σχέση με τη φορολογία των καταθέσεων δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα από το Συμβούλιο. Ήταν μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαμε κάνει στα πλαίσια της νέας εντολής μας. Δυστυχώς εκεί είμαστε. Και το θέμα είναι να προχωρήσετε γρήγορα και με αποφασιστικότητα, αλλιώς θα τσακωθούμε σε εισαγωγικά. Λοιπόν, ανά πέντε λεπτά θα προχωρήσουν οι ερωτήσεις γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Αν έχετε τέσσερα λεπτά ερώτηση θα έχετε ένα λεπτό στην απάντηση. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Πρώτος θα θέσει ερώτηση ο Ζωάν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θέλω να σας καλωσορίσω. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε και να συζητήσουμε την Προεδρία σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και για άλλο ένα λόγο, αλλά ε, σταμάτησα, διστάζω λίγο, γιατί τολμήσατε να ομιλήσετε την μητρική σας γλώσσα. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, όχι γιατί καταλαβαίνω, αλλά είναι σημαντικό ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗ να τολμά να ομιλεί την γλώσσα του. Για δυόμιση λεπτά βέβαια, παρακαλώ και την επόμενη φορά να το κάνετε. Ίσως όμως εσείς επειδή ομιλείτε πιο εύκολα την αγγλική από μένα ξέρετε να ομιλείτε και στους βουλευτές. Μας είπατε πράγματα που μας ευχαριστούν. Μας είπατε ότι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο. Μας αρέσει να το ακούμε. Είπατε ότι θα μας ακούτε και αυτό μας αρέσει. Μία ερώτηση. Έχετε, ε, είστε έμπλεος καλών προθέσεων. Πολύ καλό αυτό. Ξεκινάτε μια φιλόδοξη προεδρία και έχετε δίκιο. Επειδή δεν είστε η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πετύχετε μια εξαιρετική προεδρία. Το Λουξεμβούργο τα καταφέρνει πολύ καλά. Αλλά μετά από τη συζήτηση που είχαμε στο Κοινοβούλιο εδώ και ένα περίπου μήνα για τα θέματα τα οποία καθυστερούν στο Συμβούλιο, ε, για το θέμα της ε, Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο παρουσίασε, της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, το οποίο παρουσίασε η κυρία Μπάουλς. Ε, τι θα κάνετε για να ξεμπλοκάρετε αυτά τα θέματα. Κάντε το σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι θα κερδίσετε το χρόνο που μιλήσατε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ Ζωαπόλ, λέει ο πρόεδρος. Δυστυχώς τα γαλλικά μου είναι πολύ χειρότερα από τα δικά σου αγγλικά. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση την οποία έκανες. Είναι παρατήρηση η οποία περιλαμβάνεται και στα ψηφίσματά σας. Πράγματι, έχουμε πάρα πολλά θέματα, τα οποία έχουν κολλήσει θα έλεγα, για διάφορους λόγους. Μερικές φορές μας λείπουν τα συμπεράσματα των συζητήσεων στο Συμβούλιο, μερικές φορές υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ή τις κυβερνήσεις μεταξύ τους. Νομίζω ότι δεν έχουμε όμως κάποια άλλη επιλογή από το να προσπαθήσουμε εμείς να ρυθμίσουμε κάπως το χρονισμό των συζητήσεων και όχι μόνο, προσέξτε με, όχι μόνο σε επίπεδο Προεδρίας αλλά και σε επίπεδο εικόνα. Ήδη ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό. Ήδη έχουμε μπορέσει να, να συμπυκνώσουμε ορισμένα θέματα σε επίπεδο τριμερών διαλόγων για το μήνα Ιούλιο. Ήδη προσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε παράλληλα τις συναντήσεις μας οι οποίες θα ξεκινήσουν εκ νέου στα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Νομίζω λοιπόν όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου παρουσίαση θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας τους βασικούς στόχους ε, τους οποίους επιδιώκουμε. Πάρα πολλές φορές αυτοί οι βασικοί στόχοι δεν συμφωνούν πλήρως, δεν συμπίπτουν θα έλεγα με κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις και τεχνικές οδηγίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια κάποια ιεραρχία και να δημιουργήσουμε μια διαδικασία fast track για κάποια θέματα τα οποία θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά. Αναφέρθηκα σε κάποια από αυτά στην παρουσίασή μου. Omnibus 2, MIFID. Για να μην αναφερθώ στα της Τραπεζικής Ένωσης, και να προσπαθήσουμε να μην ε, δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλα θέματα τα οποία έχουν προχωρήσει και τα οποία απλά χρειάζονται κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις. Προσπάθησα να απαντήσω α, ε, ειλικρινά. Δεν έχουμε πολλούς πόρους και εσείς δεν έχετε πάρα πολλές δυνατότητες. Σας συναντηθούν. Εγώ θα συναντώ συχνά τη Σάρων με μεγάλη χαρά για να μπορέσουμε να ε, συμπέσουν τα χρονοδιαγράμματά μας. Μοντολίν από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω κι εγώ στη μητρική μου. Ε, Ισπανικά. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω καταρχάς τον Υπουργό. Σας προσφέρω τη συνεργασία και ε, την προθυμία της ομάδας μας. Εσείς μπορεί να είστε υπουργό οικονομικών μιας μικρής χώρας, αλλά οι μικρές χώρες κάνουν σημαντικά πράγματα για την Ευρώπη και σπουδαίες προεδρίες. Εμείς επιθυμούμε, σαφώς, να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, να ξεφύγουμε από την ύφεση και να μπούμε στην ανάπτυξη. Ορισμένες από τις ειδικές συστάσεις αναχώρα ε, που σήμερα εγκρίθηκαν πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση γιατί θέλουμε και ζητούμε εδώ και καιρό να δοθεί λίγος χρόνος στις χώρες αυτές για να γίνουν αυτές οι προσαρμογές αλλά όχι με τέτοιο ριζικό και δραστικό τρόπο. Ε, ελπίζω και εσείς να μπορέσετε να ε, προωθήσετε τις επενδύσεις. Θα συνεργαστούμε στους στόχους που αναφέρετε Θέλω να σας αναφέρω δύο ζητήματα και να σας ρωτήσω και να σας ζητήσω να δώσετε μεγάλη σημασία. Γιατί πιστεύουμε ότι μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας σας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανυπόθηκη πίστη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική οδηγία. Έχουμε ε, ολοκληρώσει τους τριμερείς διαλόγους με συμφωνίες. Αυτή τη στιγμή εκρεμεί μόνο μια διαφορά ανάμεσα σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και έχει να κάνει με τη διαδικασία υλοποίησης της οδηγίας. Ε, σας ε, συνιστώ θερμά να είστε σε διάλογο πολύ στενό με την πρόεδρο της Επιτροπής μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας μάλιστα. Εκρεμεί αυτή η μεταρρύθμιση και ε, που απομένει μια τελική όθηση για να ολοκληρωθεί. Και νομίζω ότι είναι στο χέρι σας να το πετύχετε αυτό. Και ένα άλλο που σας παρακαλώ να το κοιτάξετε πολύ προσωπικά γιατί ε, κάλλιστα μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ και να ολοκληρωθεί και στη δική σας θητεία, στη δική μας θητεία, είναι ο ανταγωνισμός και οι ε, δράσεις και οι προσφυγές ε, για να αξιώνει κανείς αποζημίωση σε περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Σας παρακαλώ να τα προσέξετε αυτά, να τα προωθήσετε και αυτό θα συνεισφέρει στο να θευθεί και με επιτυχία η ε, Προεδρία σας και να έχει αυτά αποτελέσματα. Ναι, Αντολίν, σε ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σου. Uh, ε, γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα νομοθετήματα ε, και έχω ενημερωθεί ότι είναι στο τελικό στάδιο και πραγματικά το συντομότερο θα ασχοληθούμε και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα. Και αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να πω ισχύει και για άλλα θέματα και για άλλες πρωτοβουλίες όπου υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα πρότεινα σε στενή συνεργασία βεβαίως αν χρειάζεται και με τη Σάρων ε, προσωπικά ε, αλλιώς ε, να έχουμε και ένα μέλος η Μίγκλε είναι εδώ στις Βρυξέλλες, είναι στη διάθεσή σας από την Προεδρία για αυτά τα τεχνικά ζητήματα, τα τεχνικά και τους κανονισμούς που είμαστε συνομοθέτες ας τα ολοκληρώσουμε. Μπορεί να μην μείνουν όλοι ικανοποιημένοι, να μην είναι το απάβγασμα της τελειότητας αυτό το αποτέλεσμα, αλλά καμιά φορά είναι πιο σημαντικό να επιτύχεις ένα αποτέλεσμα και ας μην είναι τέλειο. Δηλαδή, αν το τέλειο το πετύχουμε σε δύο χρόνια, ας πάρουμε μια απόφαση σήμερα και αναθεωρούμε σε δύο χρόνια. Ε, παρακαλώ ε, να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό το συντομότερο για τεχνικά ζητήματα που είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας και έχετε απολύτως δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που δεν πρέπει να λησμονούμε. Ορισμένα είναι πραγματικά σημαντικά για τους καταναλωτές, για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες που χρειάζονται την προσοχή μας και τη φροντίδα μας. Ευχαριστώ. Για τις υποθήκες το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, αν υπάρχουν ερωτήσεις, για το πώς θα εφαρμοστεί να συμφωνήσουμε. Αν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, ας απαντηθούν. Συμφωνήστε να υπάρξει ένα άρθρο που να ορίζει ότι τα κράτη-μέλη θα δίνουν κάποια περισσότερη πληροφόρηση. Δεν είναι και τραγικό αυτό που ζητάμε. Ας προχωρήσουμε τώρα στους φιλελευθέρους όλες Σμιτ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλωσορίζω τον Υπουργό Οικονομικών. Ήταν μεγάλη χαρά, πολύ ενδιαφέρον που σας ακούσαμε οι βαλτικές χώρες, η Λιθουανία. Ανάμεσα στις βαλτικές χώρες η Λιθουανία ήταν η πρώτη ε, που επισκέφθηκα μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Είσαστε γειτονική χώρα και έχουμε στενές σχέσεις. Είναι πολύ καλό που σας βλέπουμε εδώ και δείχνει ότι πόσο, πόσο μπορεί να αλλάξει η ιστορία. Ε, Τραπεζική Ένωση. Είχαμε τον κύριο Ντράγκη εχθές εδώ. Είμαι, φοβούμε κάπως ότι αν όλες οι χώρες, 28 τώρα, ε, προσχωρήσουν στην Τραπεζική Ένωση θα υπάρξει πρόβλημα για τις τράπεζες εκτός και τις χώρες εκτός ευρώ έχετε και στη χώρα σας πολλές σουηδικές τράπεζες και η Σουηδία είναι εκτός της Ευρωζώνης και εσείς είσαστε επίσης εκτός Ευρωζώνης. Αν μία από αυτές τις χώρες δεν προσχωρήσει στην τραπεζική όνεση, αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα βεβαίως. Θα στεθεροποιηθεί η Ευρωζώνη και οι χώρες της Ευρωζώνης και οι τράπεζες της Ευρωζώνης, αλλά θα δημιουργηθούν προβλήματα για τους άλλους. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Σχετικά με αυτές τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Προσπάθησα σήμερα να διαβάσω μερικές από αυτές. Οι συστάσεις για τη δική μου χώρα ελπίζω η κυβέρνηση να ακούει, αλλά δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Είδα τις συστάσεις για τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, όπου γίνεται λόγος για μισθούς, ε, ρομίστια. Ε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό στην Γερμανία ε, και πώς ε, αυτό το θεωρείτε εντός της Ευρωζώνης. Η εφαρμογή των συστάσεων γίνεται, πραγματοποιείται. Είναι το τελευταίο μου σχόλιο αναφέρεται στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων που αναφέρεται. Εάν θα ανοίξετε αυτό το φάκελο, θα ανοίξετε ίσως και την, οδηγία αποζημίωσης επενδυτών, γιατί αυτό είναι κάτι που λιμνάζει που, ε, και, εγώ θα φύγω από το Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. I in Θυμάμαι τη συνάντησή μας στο Βίλνιους μαζί με τους συναδέλφους σας της Άλντε Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε εκεί. Σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση, σχετικά με την τραπεζική όνεση, ένωση, είναι ένα πρόβλημα βεβαίως ε, που έχουμε και εμείς. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης για το θέμα της ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών. Είναι από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε επίσης και για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Θα έχουμε πάντοτε καταστάσεις όπου μία χώρα ε, είναι η χώρα που υποδέχεται και η άλλη η χώρα αποστολέας αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο και για να μην αθίξουμε τους φορολογούμενους οι οποίοι είναι σε αυτή τη σχέση. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω σχετικά με την κατάσταση της Λιθουανίας, διότι ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΙΝΑ βεβαίως μπορώ να αλλάξω καπέλο για λίγα δευτερόλεπτα. Ε, Βεβαίω και η Λιθουανία θα προσχωρήσει στην Τραπεζική Ένωση όταν ε, ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Αυτό θα συμβεί στην πραγματικότητα και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα ισχύσει. Και βεβαίως θα συμμετάσχουμε και πάλι τώρα αλλάζω καπέλο θα συμμετάσχουμε σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, ένας άλλος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Νομίζω ότι θα βρούμε λύσεις. Δεν, δεν είναι πολύ ε, απλές, αλλά τα θέματα αυτά θα λυθούν. Τώρα όσον αφορά ε, τις συστάσεις ειδικέ αναχώρα και τη μέτρησή του. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι δεν μπορούν να μετρηθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτές οι συστάσεις είναι συστάσεις για τις χώρες, για κυρίαρχες χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή της επικουρικότητας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική και πρέπει κάθε χώρα να κάνει το καθήκον της, τα μαθήματά της, με τον τρόπο που είναι καλύτερος για το λαό αυτής της χώρας. Ε, και που γνωρίζει καλύτερα η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως, ε, η αποτελεσματικότητα αυτών των συστάσεων και το γεγονός ότι δεν είναι συγκεκριμένες, νομίζω ότι είναι μια ε, τάση δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα το τέταρτο εξάμεινο, αλλά είναι καλή η κατεύθυνση σχετικά με την, ε, ε, για το καθεστώς αποζημίωσης των επενδυτών ε, σχετίζεται με τις ιδέες που θα έχουμε για το DGS για την εγγύηση των καταθέσεων ε, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για το θέμα της αποζημίωσης των επενδυτών, για να δούμε τι θα έχουμε στο σύστημα εγγύησης των καταθετών. Μετά ε, τα πράγματα θα προχωρήσουν ομαλά και θα δούμε πώς θα δράσουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω τώρα από πλευράς Πρασίνων το λόγο θα πάρει ο Πολβίσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενώνω και εγώ τη φωνή μου με τους συναδέλφους μου, Υπουργέ, για να σας καλωσορίσω εδώ και να σας ευχηθώ μια προεδρία, αν όχι ησυχή, ε, τουλάχιστον αποτελεσματική. Ακούσατε και τους συναδέλφους. Μπορεί να διαφέρουν ε, οι απόψεις και εκτιμήσεις από συνάδελφο σε συνάδελφο και είναι επόμενο αυτό και φυσιολογικό, ε, για τα θέματα. Συμφωνούμε όμως όλοι ως προς την εμπλοκή και την ατονία που παρατηρείτε ε, σε κάποια θέματα, την ακινησία. Είπατε εσείς ότι έχετε την πρόθεση και με τρόπο θελησιοκρατικό να τα προωθήσετε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα θέματα αυτά δεν είναι καθόλου ε, ανώδυνα, είναι, δηλαδή ισονοσημασίας, ε, είναι ε, βοηθούν για τη διάρθρωση μιας καλύτερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Είναι η Τραπεζική Ένωση, στην οποία αναφερθήκατε, ιδιαίτερα ως προς το σύστημα επίλυσης ε, των διαφορών της εγγύηση των καταθέσεων, είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, είναι όλο το ζήτημα το αχανές της αμοιβιοποίησης των χρεών, όλα αυτά τα ε, θέματα σήμερα έχουν οδηγηθεί σε εμπλοκή. Και θα ήθελα να σας ερωτήσω, να μας πείτε την άποψή σας από αυτό, αφού έχετε την πρόθεση, λέτε, να τα προωθήσετε. Εσείς ε, πού βλέπετε την εμπλοκή, δηλαδή η λύση από πού θα δοθεί. Ο κόμπος που βρίσκεται, δεν είναι μόνο τεχνικά τα ζητήματα που υπάρχουν και πολλά, ούτε χρονικά και τέτοια υπάρχουν, χρονοδιαγράμματος δηλαδή. Ε, αλλά υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Και αν ναι, πού ε, αυτά στο Συμβούλιο, στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στα διάφορα συμφέροντα κρατών μελών. να πιστέψουμε την ανάλυση και την ιδέα που προωθούν μερικοί ότι η γερμανική κυβέρνηση μπλοκάρει ουσιαστικά. Το ακούτε αυτό το επιχείρημα. Ε, τι πιστεύετε γι' αυτό. Και για να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση του Ζανπόλ Πολ Γκοζές προηγουμένως. προτίθεστε να κάνετε και με ποιο τρόπο θα προχωρήσετε. Θα βασιστείτε βεβαίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και με χαρά εμείς να σας βοηθήσουμε. Αλλά πώ θα έρθει, από πού θα έρθει η απεμπλοκή όλων αυτών των ζητημάτων για να μπορέσει να εκφραστεί αυτός ο βολονταρισμός. Ε, ποια είναι η νέα ευκαιρία τώρα ε, που θα επιτρέψει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είναι οι γερμανικές εκλογές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και έκβασης. Έχουμε και αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αυτή την ημερομηνία. Για εσά είναι σημαντική. Δεν σταματώ εδώ. Τώρα θα απαντήσει σύντομα, λέει η κυρία Μπόλ. Θα προσπαθήσω. Ζαν Πολ, μα τα λες με τέτοια ακρίβεια. Έχει ταυτοποιήσει με ακρίβεια όλους εκείνους τους παράγοντες που καμιά φορά εμποδίζουν την πρόοδο. Σε πολύ διαφορετικά θέματα, όντω, ανέφερε από το FTT ε, το φόρο επί των πιστωτικών συναλλαγών, το Ταμείο Εξυγίανσης. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και κρατών μελών και όχι μόνο. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ ε, των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάμεσα και στο εσωτερικό πολλές φορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καμιά φορά έχουμε ανεπαρκή πρωτοβουλία και άλλοτε υπερβάλλοντα ζήλο χρέος και καθήκον της ε, Λιθουανικής Προεδρίας είναι να είμαστε ειλικρινείς διαμεσολαβητές για να σφυριλατούμε συμβιβασμό. Ε, εγώ ε, θα συναντώ τους ενεχομένους, θα συζητώ, θα τους κοιτώ στα μάτια, θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Το κάνω και με τους συναδέλφους υπουργούς με τους οποίους έχω συναντηθεί με τους ομολόγους μου πάρα πολλές φορές. Ε, και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω συναντηθεί με πολλούς από εσάς στο παρελθόν. Με άλλους όχι. Και δεν υπάρχει πρόβλημα να συναντηθώ στο μέλλον. Και σε αυτές τις συζητήσεις πιστεύω ότι θα εντοπίσουμε ακριβώς ε, τα εμπόδια. Ε, βεβαίως καμιά φορά υπάρχει και ο πολιτικός κύκλος που υπαγορεύει το χρονισμό. Ε, πολιτικοί είμαστε. Γνωρίζουμε ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν πολιτικά ημερολόγια καμιά φορά που επηρεάζουν τα πράγματα. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, δεν υπάρχει καμιά πανάκια, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Ο Γιώργεν Κλούτε τώρα από την Γκουε. Ευχαριστώ, Σάρον. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω θερμότατα εξ ονόματος της ομάδας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Εδώ είμαι. <laughs> Ich Είναι σημαντικό πιστεύω αυτά που έχετε καταρτήσει ως κατάλογο να τα φέρετε και σε πέρας πριν λήξει η θητεία. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα θέμα το οποίο ήδη απαντήσατε και αυτό είναι την ε, οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών. Είπατε ότι θέλετε να το βάλετε στην ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι συγκητής για αυτό το θέμα και είχαμε αποτανθεί και σε εσά και καλωσορίζω αυτή τη δήλωσή σας ότι το έχετε εντάξει στον κατάλογο προτεραιοτήτων. Θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Σήμερα κάναμε εδώ την πρώτη συζήτηση και φιλοδοξούμε να το διεκπαιρεώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι υπάρχουν και μεγάλες πιθανότητες. Έχω όμως και ένα άλλο σχόλιο να κάνω σχετικό με αυτό εγώ είμαι Γερμανός ε, και να πω αυτό που είπε και όλος Σμιτ και να ρωτήσω. Έχετε κάνει συστάσεις ειδικέ χώρα. Τι κάνουν οι χώρες. Η Γερμανία και πέρυσι και φέτος ε, πήρε πολύ σαφές συστάσεις. Ε, προσωπικά λυπάμαι που στη Γερμανία αυτό δεν υιοθετείται, γιατί θα ήταν σημαντικό για να ε, ξεπεραστεί η κρίση και είπατε ότι είναι σχόλια, είναι συστάσεις, σημειώσεις, υποδείξεις, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και την κυριαρχία των κρατών και την αρχή της επικουρικότητας. Ωραία είναι όλα αυτά και τυπικά πάρα πολύ σωστά. Από την άλλη όμως τις χώρες που έχουν ελλείμματα επεμβαίνεται σε μεγάλο βαθμό στην κυριαρχία τους και αυτό ε, είναι ανισότητα και αυτή η ανισότητα είναι όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνεργασία και ε, στην αλληλεπίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ η εκτίμησή σας. Ευχαριστώ. Ja, uh, Jürgen. στα γερμανικά. Ευχαριστώ Γιώργεν. Δυστυχώς τα γερμανικά <laughs> δεν είναι η ειδικότητα μου, ούτε η γλώσσα εργασίας. Αγγλικά μιλάμε συνήθως. Και θα απαντήσω στα αγγλικά, μέχρι εδώ τα γερμανικά. Η οδηγία για τις πληρωμές έχει προχωρήσει αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει τις δικές της προτάσεις και όλα τα στοιχεία τα οποία έχει. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση καταρχάς γενικότερη γύρω από αυτό στο Συμβούλιο. Η πρώτη ομάδα εργασίας για την οδηγία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς προβλέπεται να συνεδριάσει τον μήνα Σεπτέμβριο. Υπάρχουν δυνατότητες δηλαδή για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Η ερώτησή σας τώρα για τις συστάσεις για συγκεκριμένες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οι συστάσεις αυτές πριν ένα χρόνο δεν υπήρχαν ουσιαστικά. Τώρα έχουμε τα μέσα που θα τις δημιουργήσουμε. Έχουμε επίσης και τις διαδικασίες αντιμετώπισης ε, των μακροοικονομικών ανισοτήτων. Θα περάσουμε επίσης και στην καταγραφή των δικτών των κοινωνικο-οικονομικών από το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το σύστημα θα λειτουργήσει σωστά γιατί απαιτεί χρόνο και πολλή ενέργεια. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχουμε προχωρήσει όχι με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά έχουμε καταστήσει πιο συγκεκριμένες τις συστάσεις αυτές προς τις διάφορες χώρες και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε και σε επίπεδο αριθμών, αν θέλετε και να μην μείνουμε μόνο σε επίπεδο θεωρητικό, ακαδημαϊκό, σε επίπεδο ιδεών για το πώς θα αλλάξει το συνταξιοδοτικό, το πώς θα αλλάξει το εργατικό δίκαιο. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία θα σημειωθεί πρόοδος. Το υπόσχομαι. Υπόσχομαι επίσης ότι θα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτό να μην οδηγήσει στην αύξηση του διοικητικού γραφειοκρατικού βάρους σε επίπεδο το οποίο θα είναι ε, ε, ο λίγων ευφυές. Θα πρέπει να υπάρξουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις του ταχύτερο δυνατόν. θα προχωρήσουμε την επιδίωξη παράλληλα διαφορετικών στόχων και θα δούμε το φθινόπωρο πώς η αξιολόγηση εξάντε των προϋπολογισμών θα προχωρήσει και θα έχουμε συλλέξει στοιχεία για το πώς να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πλέον. Ευχαριστώ. Η ε, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Εδώ είμαι. Καλώς όρισατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην Προεδρία σας. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι επιζητείτε τη συνεργασία και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις ε, φιλονικίες και τους διαξυφισμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά θέλει να δει αποτελέσματα και συμφωνώ με αυτό που είπατε και με χαρά να συνεργαστούμε. Ε, σύνθημα της ε, Προεδρίας σας είναι να προχωρήσετε σε αποτελέσματα, είπατε, και για την Τραπεζική Ένωση και ελπίζω ε, να το προωθήσετε και όλα αυτά τα ζητήματα των τραπεζών. Βλέπω ότι αναφέρεται μια σειρά ζητημάτων της Τραπεζικής Ένωσης, όπου εργάζεστε σκληρά. Έχω ε, τις εξής ερωτήσεις. Για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό Έχουμε προγραμματίσει στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο να ψηφιστεί. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα έτσι χρονική για το πότε θα λυθεί αυτό οριστικά, να περάσει από την Ολομέλεια το Σεπτέμβριο στο Συμβούλιο, ε, πότε θα ε, τεθεί σε λειτουργία. Και το δεύτερο, το ε, ενίο μηχανισμό εξυγίανσης, θα κάνει μια πρόταση ο Επίτροπος Μπαρνιέ, αύριο, ορισμένες χώρες δηλώνουν ότι αυτό προϋποθέτει αναθεώρηση συνθήκης. Ακούω διάφορες φήμες ε, στους διαδρόμους ότι ε, θα προβάλλουν δυσκολίες ορισμένες χώρες. Ποια είναι η πρόθεση της Λιθουανικής Προεδρίας. Για να υπάρξει ένας ενιαίος μηχανισμός, δηλαδή καθάριση χρειάζεται αναθεώρηση συνθήκης ή όχι. Και για τη φοροδιαφυγή ε, και τη φορολόγηση ε, των εσόδων από εκεί. Είπατε ότι είναι κλεμμένα τα χρήματα αυτά και συμφωνώ. Αλλά το, όταν πρόκειται για το CCTB που είναι η ενιαία ολοκληρωμένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις, δεν βλέπω πολύ μεγάλη φιλοδοξία στο Συμβούλιο. Γιατί πια είναι τόσο δύσκολο τεχνικά να καταλήξετε σε μια οριστική θέση ή μήπω υπάρχει πολιτική απροθυμία και πάλι για να προωθηθεί. Εγώ ήμουν εδώ η συγκήτρια και είναι ένα μέσο που μπορεί να μας βοηθήσει για να αποφύγουμε αυτή την επιθετική ε, προσφορά φοροδιαφυγής. Α, δεν μίλησε η Μαριάννα 8 λεπτά, το ρολόι είχε πρόβλημα. Ναι. Απαντήστε παρακαλώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ Μαριάν. Σημαντικά τα ερωτήματα αυτά. Ο νέος ε, εποπτικός μηχανισμός είναι ε, εξαιρετικά σημαντικός και ε, προσωπικά θα επιθυμούσα και εγώ και το Συμβούλιο να ε, ψηφιστεί το συντομότερο. Και η Γερμανική Βουλή ε, που επρόκειτο να ψηφίσει τώρα υπερψήφισε ήδη. Το πρόβλημα είναι ότι τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά ε, την ψήφιση και τη δημοσίευση στην ε, επίσημη εφημερίδα. Δηλαδή όσο αργότερα το ψηφίσετε τόσο αργότερα θα υλοποιηθεί. Ε, είχε προγραμματιστεί για τα μέσα του 2014. Τώρα μπορεί να πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2014. Αν μου επιτρέπετε να σας απευθύνω μία έκκληση, σας παρακαλώ. Ψηφίστε το το συντομότερο. Εγώ δεν μπορώ να σας προτείνω πώς θα κανονίσετε τις εργασίες σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι στις δυνάμεις μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για τον νέο μηχανισμό εξυγίασης, ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε ότι θα κάνει μια πρόταση αύριο. Οι προτάσεις αυτές θα συνάδουν ε, με τις κείμενες συνθήκες. Προς το παρόν, για το δικό μας εξάμεινο δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ε, θα πρέπει να κινηθούμε εντός των κειμένων ε, ε, συνθήκων. Και όσο γίνεται θα το κάνουμε και θα δείξει το μέλλον. Την πρόταση δεν την έχω δει. Ας περιμένουμε να δούμε. Και το τελευταίο που με ρωτήσετε για το CCTB, την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις, η μοίρα αυτού του θέματος που εκρεμεί επιτάπητος εδώ και καιρό, για μια δεκαετία αν δεν απατώμε, είναι ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Ε, ακούω ότι υπάρχουν μερικές ιδέες τώρα να διαχωριστούν ορισμένα στοιχεία από αυτό το φάκελο, έτσι ώστε να μπουν στην άκρη τα πιο επίμαχα σημεία και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τα άλλα που είναι πιο συνενετικά. Ε, στα οποία συμφωνούν σχεδόν όλοι. Αυτό όμως χρειάζεται τεχνική δουλειά και στη φορολογία, ιδιαίτερα στην άμεση φορολογία, όπου δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοχή χρειάζεται εκεί. Θα πρέπει να ακούσουμε όλους τους ενδιαφερομένους και χρειάζεται εκεί ομοφωνία μεταξύ υπουργών και κυβερνήσεων και πολιτική υποστήριξη φυσικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσουμε σε αυτό το δρόμο και θα δούμε τι είναι εφικτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολιτική υποστήριξη είχατε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το CCCTB. Πριν από μια πενταετία έκανα την έκθεσή μου για τη φορολογία. Ε, το ξέρω ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Θυμάμαι ότι ρώτησα, ζήτησα κάτι από τον Αντόλφο να με ενημερώσει, λέει ναι ξέρω τι θέλεις και μου στείλε 2.000 σελίδες. Ε, το ξέρω ότι είναι περίπλοκο. Η Μαριάν έχει κάνει όμως πολύ καλή δουλειά ε, από πλευρά του Κοινοβουλίου. Για τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό, το SSM, θα ψηφίσουμε ε, όταν συμφωνήσουμε για τα θέματα λογοδοσίας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την οποία είχαμε άλλη μακρά συνεδρίαση σήμερα. Θα πρέπει επίσης, και είναι απαραίτητο να λυθεί αυτό, για να υπάρχει μια ασφάλεια για τα κράτη-μέλη, τα κοινοβούλια, να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυρία Κράτσα, παρακαλώ, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Υπουργέ, θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα, την ελληνική. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησα και την παρουσίαση των προτάσεων και τις απαντήσεις που δώσατε στους συναδέλφους μου. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στο πρόβλημα της χρηματοδότησης της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας και ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρειαστούμε μέχρι το 2020 1,5 με 2-3 ευρώ. Και ήδη έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού ταμείου ε, στο οποίο για να διευκολύνει τις ε, ε, επενδύσεις των θεσμικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ήθελα να ρωτήσω τι θέση θα έχει αυτό το θέμα στην ε, Λιθουανική ε, Προεδρία. Αν ε, έχετε, το έχετε ήδη στις προτεραιότητές σας, πώς κρίνετε την πρόταση ήδη που έχει κατατεθεί, αν ξέρετε τις αντιδράσεις στο Συμβούλιο, στην αγορά, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε και τα πραγματικά εργαλεία αλλά και την ελπίδα στους επενδυτές ότι θα βρεθούν, θα βρεθούν διέξοδοι και δυνατότητες επενδύσεων σε μακροπρόθεσμα σχέδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν, Ρόδη, για την ερώτησή σου για αυτό στις ερωτήσεις. Πρόκειται για μια πολύπλευρη ερώτηση θα έλεγα. Βεβαίως η πηγή χρηματοδότησης είναι σημαντική, αλλά από μόνες τους δεν λύνουν το πρόβλημα αυτές οι πηγές. Χρειάζονται μέσα εργαλεία, όπως σωστά αναφέρατε, χρειάζονται, χρειάζεται επίσης ένα κλίμα επενδυτικό στις χώρες, σε πάρα πολλές χώρες. Στη δική μου χώρα στις γείτονες μας, στην Λετωνία, μία από τις μεθόδους για να βελτιωθεί το κλίμα το επενδυτικό είναι η προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Είναι ένα πραγματικό βήμα προόδου για την βελτίωση του κλίματος του επενδυτικού για να έρθουν ιδιωτικές επενδύσεις. Μιλούσαμε για δημόσια κονδύλια και νομίζω ότι τα δημόσια κονδύλια στην Ευρώπη είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης και θα έπρεπε ε, να χρησιμοποιηθεί ε, με σόφρονα τρόπο. Έχουμε πολλαπλές πρωτοβουλίες. Έχουμε την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων που συζητήθηκε στην συνάντηση των αρχικών κρατών και στο επίπεδο του ΕΚΟΦΗΝ σήμερα. Αυτά τα θέματα ίσως να μπουν στην ατζέντα του άτυπου ΕΚΟΦΗΝ που θα έχουμε στο Βίλνιους ε, και ε, θα ήθελα να καλέσω τη Σάρον και μέλη της Επιτροπής σας να συμμετάσχουν ε, σε αυτήν τη σημαντική συνάντηση. Είναι πολύ καλή παράδοση μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύο φορές το χρόνο να συμμετέχουν στα άτυπα συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ. Νομίζω ότι είστε προστιθέμενη αξία στη συζήτηση των θεμάτων αυτών. Μια άλλη πηγή είναι απλώς ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός και έχουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που ξέρουμε που βρισκόμαστε. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να επιληθεί, να επιληθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Είμαι επίσης υπεύθυνο για την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχή και θα έχουμε τον Νοέμβριο συνάντηση των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για τη συνοχή. Αυτό είναι ένα άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσατε να συμμετάσχετε. Ίσως δεν είναι πολύ ενδιαφέρον για σας, είναι πιο ενδιαφέρον για την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, αλλά θα μπορούσατε να ξανάρθετε στο Βίλνιος και θα συζητήσουμε ε, πώς οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί και τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο με χορηγήσεις αλλά ε, για τα σχήματα, για την αρχιτεκτονική των διαφόρων χρηματοδοτήσεων, για την καλύτερη χρήση των χρημάτων. Νομίζω ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα. Επίσης έχουμε πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την χρηματοδότηση και περιμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για τα θέματα αυτά, δηλαδή την μη τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Είναι πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η οικονομία μας κυρίως χρηματοδοτείται από τις τράπεζες. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων προέρχεται κατά 80% από τράπεζες. Αυτό είναι διαφορετικό στην Αμερική, όπου μόνο 20-25% 80% προέρχεται από τράπεζες και το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία και άλλα μέσα αυτού του είδους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας ανοιχτός τομέας όπου χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα, να συζητήσουμε. Νομίζω στο συνεδριάσεις της ΕΚΟΦΗΝ θα επανέλθουμε στις ιδέες αυτές. Ε, με πολύ χαρά θα συζητούσα και τις ιδέες αυτές μαζί σας επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Σίμων από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Υπουργέ, για την τοποθέτησή σας. Εδώ είμαι. Για το, τις προγραμματικές σας δηλώσεις για το πρόγραμμα εργασίας. Εγώ είμαι εισηγητής για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και χαίρομαι πάρα πολύ για την προσοχή που δίνετε ε, σε πρώτη ανάγνωση ψηφίστηκε πριν από μια 1,5 χρόνο αυτό το θέμα. Χαίρομαι που θα αφοσιωθείτε. Ξέρουμε ότι το παράθυρο αυτό της ευκαιρίας είναι μικρό και οι πόροι όλων των ενεχομένων περιορισμένοι. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι θέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ύψος των ταμείων, είναι τελείω αποκλίνουσες. Αλλά ε, στη δική σας Προεδρία βλέπω πραγματικά μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας από κοινού να φέρουμε σε πέρας δύο πράγματα που πρέπει από κοινού να έρθουν σε πέρας. Είναι το Ταμείο Εξυγίανσης και Ανάκαμψης, αυτός ο μηχανισμός, και το άλλο είναι η εγγύηση των καταθέσεων με ένα άλλο ταμείο, ξεχωριστό. Γιατί το Συμβούλιο συνδέει το ύψος των πόρων των δύο ταμείων. Συμφωνώ πολύ τους μαζί σας όταν λέτε ότι θα πρέπει να συνδέσουμε, να συνδυάσουμε αυτά τα θέματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά το ύψος της πρικοδότησης ε, για τα δύο ταμεία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ακόμα και αν είναι από τη δική μας άποψη δύο διαφορετικά ταμεία αυτά. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα σημεία που πρέπει να κάνουμε χωριστά τις διαπραγματεύσεις. Και σας ερωτώ, θέλετε να κάνετε παράλληλα τις διαπραγματεύσεις. Τι εννοείτε? Ότι ο τριμερής διάλογος θα γίνεται συνολικά από κοινού ή θα έχουμε τελείως ξεχωριστές τριμερείς διαπραγματεύσεις. Εμείς αυτό θα το κολοσορίζαμε πέρα από την πρικοδότηση των ταμείων και το πραγματικό ποσό. Ε, τελικά δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουμε ούτε εσείς ούτε εμείς. Έχουμε όμως νομίζω καλές πιθανότητες ε, στη δική σας Προεδρία να τα κλείσουμε αυτά τα θέματα αν πραγματικά αρχίσουμε το Σεπτέμβριο την ουσιαστική δουλειά. Ναι. Πέτερ, ευχαριστώ στα γερμανικά, αλλά μέχρι εδώ τα γερμανικά θα συνεχίσω την απάντησή μου στα αγγλικά. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι και τα BRD και το DGS είναι δύο θέματα τα οποία συνδέονται στενά μεταξύ τους. Συνδέονται όχι μόνο λόγω του μεγέθους των ταμείων, υπάρχουν και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες και δεν θα μπορούσα τώρα και ζητώ συγγνώμη να μπω σε λεπτομέρειες. Καλό είναι όλες οι πλευρές να ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου όταν είμαστε προετοιμασμένοι μπορούμε να συζητήσουμε εναλλακτικέ, μπορούμε να συζητήσουμε την επιλογή την οποία έχουμε να κάνουμε. Αυτά για το τεχνικό κομμάτι, αλλά πολιτικά όπως είπα στην εισαγωγική μου παρατήρηση ξεκινάμε για τον BRD τον τριμερή διάλογο αύριο 10 Ιουλίου και το σχήμα της, ε, ε, των εγγυήσεων των καταθέσεων θα συζητηθεί σε μια πρώτη φάση σε ένα βασικό επίπεδο και έχει, θα γίνει συζήτηση σε βασικό επίπεδο γιατί χρονολογικά έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Οι τριμερείς διάλογοι για τις εγγυήσεις των καταθέσεων προβλέπονται επίσης για τις αρχές ε, ε, του φθινοπόρου. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Πάντως το ταχύτερο δυνατόν, μόλις βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος. Έχουμε κάποιες πρώτες ιδέες για το τι πρέπει να κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτόν τον τριμερή διάλογο και γι' αυτό θα ζητήσω και από δική σας πλευρά να συντονιστούμε χρονικά και με τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ξαφνικά κάποιος άλλος έχει μια ευνίδια επιθυμία να θέσει ερώτηση. Όχι, σας ευχαριστούμε. Τελειώσαμε νωρίτερα. Σας περιμένουμε να ξανάρθετε και να μας πείτε πώς έχουν προχωρήσει και ολοκληρωθεί όλα τα προβλήματα και οι φάκελοι που έχετε μπροστά σας. And I can just remind us... Θα ήθελα απλώ να θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι 5η 5 Σεπτεμβρίου 9 η ώρα το πρωί. And have a good holiday. Also for the chair.